Good afternoon, colleagues. My apologies for being late. Ε, συγγνώμη για την καθυστέρηση, συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε. ενημερωθούμε για τον τριμερή διάλογο, ο οποίος έγινε στις 29 Νοεμβρίου. Θα μας ενημερώσει λοιπόν η συγγήτρια για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ αγαπητέ Κλοντ, θα είμαι σύντομη. Πρόκειται για ε, πλαστές προξενικές θεωρήσεις οι οποίες κυκλοφορούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην βάση των προτάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων από το 2015 έχει αποφασίσει να βάλει νέα τεχνικά χαρακτηριστικά στα έντυπα για τις προξενικές θεωρήσεις. Ήδη από τον Φεβρουάριο του προηγούμενου χρόνου έγινε εγκρίθηκε η διαπραγματευτική εντολή και άρχισε από τις 30 Μαΐου. Στο μεταξύ έχει περάσει κάποιο διάστημα βέβαια. Στις 29 Νοεμβρίου έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος, στον οποίο τριμερή διάλογο που εξελίχθηκε πολύ επικοδομητικά, προέκυψαν δύο συμπεράσματα, τα οποία βέβαια πρέπει ακόμα να διασαφηθούν. Το ένα που νομίζω είναι και το σημαντικότερο, πρόκειται για το θέμα εάν η Ιρλανδία θα συνεχίσει να συμμετέχει στο κοινό σύστημα των θεωρήσεων και επομένω να εφαρμόζει τον κανονισμό. Εδώ μεταξύ Κομισιόν και Συμβουλίου υπάρχουν διαφορετικές νομικές τοποθετήσεις σχετικά με το πώς θα γίνει αυτό. Αυτές οι νομικές προσεκίσεις εξακολουθούν να υπάρχουν και εμείς ως Κοινοβούλιο αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να παίξουμε έναν μεσολαβητικό ρόλο όλα τα θεσμικά όργανα επιθυμούν πάντως να, παραμείνει, να γίνει μάλλον τμήμα του κανονισμού η, Ιρλανδία. Δεύτερο, διάρκεια της μεταβατικής περίοδου και για, για πόσο διάστημα κόπη θα ισχύουν τα ε, έντυπα ευρωξενικών θεωρήσεων που υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα στις χώρες μέλη. Πάντως υπάρχει η πεποίθηση ότι μέσα στα, στη διάρκεια τη Μαλτέζικη Προεδρία θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση για τα δύο αυτά ερωτήματα. Νομίζω λοιπόν ότι ε, δεν θα χρειαστεί και πάρα πολύ χρόνο και πάντως θα, θα προλάβουμε μέσα στη Μαλτέζικη Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Ζεράρ Πρέ, επ' Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε η συγγήτρια πρόκειται για μικρό φάκελο αλλά σημαντικό διότι πρόκειται για τον αγώνα κατά της πλαστογράφησης εγγράφων ε, προκειμένου ε, αυτών των ε, σημάτων που μπαίνουν πάνω στις προξενικές θεωρήσεις και που πλαστογραφούνται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια για την προσπάθεια που έχει καταβάλει για, για το φάκελο αυτό. Έχω συνεργαστεί κατά επανάληψη μαζί τη. Καλή συνεργασία και με τους και οδησυγητές και εύχομαι καλή επιτυχία στις προσπάθειες τη και σύντομα, διότι είναι κάτι το οποίο έχει αναλάβει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ε, με πολύ ευφυή τρόπο το χειρίζεται. Μάλιστα λοιπόν, ιδού ο έπαινος από τον σκιώδη συγητή των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Ο επόμενο τριμερής διάλογο θα είναι την επόμενη εβδομάδα που φαίνεται λέει εδώ. Θα δούμε τέλο πάντων. Ευχαριστώ. Και θα επανέλθουμε. Δέκα έως 20. Απαλλαγή 2015. Ο κύριος Γέσεκ. Α, με συγχωρείτε. Ζεράρ, εσείς τον αντικαθιστάτε, έτσι δεν είναι. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ήταν πολύ επαγγελματική η έναρξη του απογεύματος. Αν θέλετε, Γεράρ πάντως, ούτως ή άλλως τα καταφέρνετε πάντοτε θαυμάσια. Uh, merci, Président. Donc, je n'interviens pas à titre... Κύριε Πρόεδρε, δεν παρεμβαίνω προσωπικά. Αντικαθιστώ τον συνάδελφο Γέρζεκ ε, και εκπροσωπώντας ε, και την ε, ομάδα ALDE. Θα ήθελα ο εισηγητής θα σα πω τα όσα προτίμασε ο κύριο Ζέκο, γιατί δεν το είχα αναλάβει εγώ. Αρχικά λοιπόν θέλει να εκφράσει την ικανοποίηση του εισηγητή σε ό,τι αφορά την ε, μείωση του περιορισμού του ε, ορίου σφαλμάτων για τον προπολογισμό του 2015, ιδίω σε ό,τι αφορά ε, τι προκλήσει ε, τι οποίε αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Με ικανοποίηση διαπιστώνει την επαγγελματική κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού στην Ευρώπη. Επίση, ο εισηγητή θέλει να ενθαρρύνει την Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων να δώσει πιο συγκεκριμένε ε, από την άλλη πλευρά ε, ε, αιτιολογήσει για του πόρου που δόθηκαν για την υποδοχή και μετεγκατάσταση. Γιατί δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία στην έκθεση τη Γενική Διεύθυνση Home. Γι' αυτό ο εισηγητή θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει πιο, πιο πλήρη εικόνα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των πόρων. Μετά, για την απαλλαγή για τους επιμέρους οργανισμούς. Ε, ο εισηγητής ε, συγχαίρει ε, τις υπηρεσίες αυτές που αντιμετώπισε και έκτακτες περιστάσεις το 2015 και θεωρεί ότι οι πόροι έχουν αξιοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο. Όμως, ζητά από τον Frontex να μεριμνήσει τους ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική διαχείριση και πιο συγκεκριμένα εστιάζει στον Frontex, γιατί είχε υποτιμήσει το κόστος ε, της, ε, ε, των περιπολιών στη θάλασσα ύψους 1,7 δις. Υπήρχαν περιπτώσεις σκαφών που είχαν περάσει από, την, από τον κύκλο ζωής του και τελικά Ο Frontex ε, ανέκτησε μόλις με 0,6 εκατομμύρια από τα 1,4 των ε, παράτυπων αυτών πληρωμών. Ο κύριος Ζέζεκ για τη ΣΕΠΟΛ τώρα υπενθυμίζει την αρχική θέση της ομάδας μας ότι ε, η συγχώνευση ΣΕΠΟΛ και Ευρωπόλ όπως είχε προβληθεί αρχικά θα ήταν ένα σημαντικό μέτρο εξοικονόμησης χρημάτων που φτάνει συνολικά στα 17,2 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς ε, δεν ε, ε, αποφάσισε το ίδιο οι συνομοθέτες, όμως ο, ο εισηγητής υπενθυμίζει αυτά τα στοιχεία. Κλείνοντα. ο εισηγητή θεωρεί ότι εν γέννη είμαστε αντιμέτωποι με ανεπάρκεια πιστώσεων πληρωμών και με αυξημένο κόστος. δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίε στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την, τον τρόπο αντιμετώπιση τη κρίση πληρωμών και είναι σημαντικό για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό στον τομέα τη δικαιοσύνη και των ιστορικών υποθέσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Ο κύριο Ζεζέκ ε, περιμένει τι τροπολογίε των συναδέλφων από τι υπόλοιπε ομάδε για να τι συζητήσει με του χειώδει τι επόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά είχα να πω για τις απαλλαγές. Ευχαριστούμε πολύ. Προθεσμία υποβολή ε, τροπολογιών η 17η Ιανουαρίου μέχρι τις 7 το απόγευμα και προβλέπεται ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 9 Φεβρουαρίου. Πριν κλείσουμε όμως αυτό το ζήτημα, να ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις ε, για κάποια από τις 11 αυτές ε, γνωμοδοτήσεις. Μόνο εγώ ακούω θόρυβα, δεν ξέρω. Όχι από τα μέλη βέβαια. Μάλλον εγώ ακούω φωνές. Παρακαλώ, κάτι θες ε, να ρωτήσεις κάτι. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση, αν μου επιτρέπετε, λέει η κυρία Κίνιτσι. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές, την εισηγήτρια βασικά και τον κύριο Ντεπρές που την αντικατέστησε. Θέλω να τους ευχαριστήσω λοιπόν για τη δουλειά που έκανε και η οποία πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Η διαδικασία απαλλαγής είναι σημαντική γιατί αντιπροσωπεύει μια θα έλεγα ευκαιρία σύγκρισης των δημοσιονομικών επιδόσεων των εξωτερικών υπηρεσιών. Και όπως είπε και ο προηγούμενος ο συνάδελφος, τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν κάποιες πολύ δύσκολες και περίπλοκες καταστάσεις, οι οποίες μάλιστα δημιουργήθηκαν με πολύ ταχύ τρόπο, κάτω από την πίεση των τρομοκρατικού φαινομένου και του φαινομένου της ε, μαζικής μετανάστευσης, και τίθεται θέμα πλέον θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα συνεχίσουν οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν τα επόμενα χρόνια και πώς έχουν δείξει μέχρι τώρα την προσαρμοστικότητά τους σε νέες και περίπλοκες καταστάσεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπογραμμίστηκε το ίδιο πράγμα ακριβώς και από το ελεγκτικό συνέδριο, ότι δηλαδή υπάρχουν διαφορές στις επιδόσεις των διαφόρων εξωτερικών οργάνων. Και σε αυτούς τους τομείς και σε αυτούς τους οποίους έθεσε ο κύριος Ντεπρέ θα πρέπει να εμβαθύνουμε μέσω τροπολογιών και στα πλαίσια της συνάντησης των σκιωδών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επιβεβαιώσω προς την Επιτροπή μας ότι είμαι διατεθειμένη να συνεχίσω να εργάζομαι επικοδομητικά, όπως συνήθως γίνεται στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά λοιπόν τους εισηγητές και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ξέχασα να πω ότι είσαι εισηγήτρια για τους σοσιαλιστές. Έχουν πει και άλλοι σκιώδεις ε, ότι θέλουν το λόγο. Τρεις συνάδελφοι Μπόνι. Εγώ αντικαθιστώ τον σκιώδη εισηγητή μας, τον κύριο Τσεχόρσκι, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον κύριο Ντεπρέ για την παρουσίαση. Οι γνωμοδοτήσεις ε, είναι πραγματικά σχετικές και αναφέρονται στα θέματα τα οποία κατατρέχουν τις εξωτερικές υπηρεσίες εδώ και καιρό. Ευχαριστώ επίσης για την πλήρη έκθεσή του και το ελεγκτικό συνέδριο. Όλες οι εξωτερικές υπηρεσίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για μας ιδιαίτερα στα πλαίσια της διαχείρισης της κρίσης της μεταναστευτικής. Γι' αυτό υπάρχουν κάποιες αυξήσεις στον προϋπολογισμό και στο προσωπικό, αλλά με υψηλά επίπεδα ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή κοινοτική προστιθέμενη αξία. Να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα τώρα σημεία σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η ΆΣΟ θα πρέπει να είναι συμβατή η διαχείρισή της με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς και να βελτιώσει τον χρονισμό των πληρωμών. Διότι και οι σκιώδεις προπληρωμές και οι καθυστερήσεις των προκαταβολών έχουν αυξηθεί το 2015 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Για τον επόπτη της προστασίας ιδιωτικών δεδομένων ε, έχουν υπάρξει βελτιώσεις στην συνεργασία και με την Ευρωπόλ και στα πλαίσια ε, της διαδικασίας του νέου μέσου ελέγχου. Ήταν νομίζω ε, έφτασε ο καιρός για να υπογραφεί η τελική συμφωνία ανάμεσα στο Frontex και την Πολωνία για την έδρα της υπηρεσίας αυτής. Απαιτείται βεβαιότητα για την λειτουργία της έτσι ώστε να καταστεί ένα ικανό μέσο για την μετανάστευση. Τώρα, συνεργασία σε ΠΟΛ και ΕΡΟΠΟΛ. Έχουμε αμφιβολίες για τη συγχώνευσή τους. Ε, θα πρέπει να παραμείνουν ξεχωριστές γιατί έχουν διαφορετικές αποδιότητες. Despite of new challenges and Νομίζω ότι θα πρέπει και η τελευταία υπηρεσία να προσαρμοστεί καλύτερα στις νέες αποστολές τις οποίες έχει αναλάβει και στα πλαίσια της συζήτησης θα προσπαθήσουμε να βρούμε λοιπόν ε, το EU lisa πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή, να ευχαριστήσω τον Ντεπρέ για την παρουσίασή του, ζητώ συγγνώμη που ήρθα καθυστερημένη. Αυτό το οποίο βρήκα σημαντικό θα έλεγα είναι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τις δαπάνες, ιδιαίτερα τα κεφάλαια τα σχετικά με την επανένταξη των Ρωμά και την εξωτερική πολιτική σε σχέση με την ε, μετανάστευση. Ε, θα ήθελα λοιπόν να εντάξουμε πολλές από τις προτάσεις ε, του συνεδρίου στις τροπολογίες τις οποίες θα κάνω, ιδιαίτερα για την πολυδιάσπαση των πιστώσεων, την απουσία ποιοτικών και όχι μόνο ποσοτικών δικτών, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει την ποιότητα των προγραμμάτων και πιο συγκεκριμένα ε, την ε, χαμηλότατη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στα πλαίσια της καταπολέμησης της βίας. Εδώ θα έλεγα το ελεγκτικό συνεδρίο κάνει σωστές παρατηρήσεις. Συμμερίζομαι τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου επίσης και για τα κονδύλια τις δαπάνες στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής γύρω από τα μεταναστευτικά θέματα. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα περιλαμβάνουν σχεδόν πάντα κάποιες συγκεκριμένες ρήτρες, σαφείς ρήτρες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όμως, ε, τα δικαιώματα αυτά δεν γίνονται πάντα σεβαστά κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Έτσι λέει το συνέδριο, δεν το λέω εγώ και αυτό ισχύει κυρίως για το Σαχάρα Μέντ, το οποίο διαχειρίζεται την μη τακτική μετανάστευση στη Λιβύη και ασχολείται με το θέμα του ελέγχου της μετανάστευσης γενικότερα στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ. Τέλος, για τους συντηρητικούς. Μακαβέη. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ ορισμένε παρατηρήσει σε ό,τι αφορά αυτού του οργανισμού. Αυτού που συνδέονται τουλάχιστον με το πεδίο αρμοδιοτήτων τη δική μα Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τι ε, δηλώσει ε, συμφερόντων, σκοπό του είναι να προλάβουν και να περιορίσουν ε, τη σύγκρουση συμφερόντων. Όλοι οι οργανισμοί, η διοίκησή του μάλλον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών των οργανισμών ε, οφείλουν ε, να ε, δημοσιεύουν τέτοιες δηλώσεις έλλειψης σύγκρουσης συμφερόντων. Και έτσι δηλώνουν ότι δεν υπάρχει τέτοια σύγκρουση συμφερόντων και είναι κάτι το οποίο υπογράφουν. Όμω θεωρώ παράλογο οι ίδιοι να δηλώνουν ότι απλώ δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Κάποιο άλλο θα πρέπει να το ελέγχει αυτό. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν δηλώσει ε, συμφερόντων, σε ποιου δηλαδή οργανισμού συμμετέχουν ω μέλη. Εμεί δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό διαφορετικά. Μετά, υπάρχει και η δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Οι διευθυντέ είναι αυτοί που συμπληρώνουν και κάποιο άλλος θα πρέπει να επαληθεύει, εάν υπάρχει ή όχι σύγκρουση συμφερόντων. Όμως, βρήκαν ένα πλαίσιο στο οποίο ουσιαστικά δηλώνει μόνο στο καθένας ε, τι είναι και τι δεν είναι. Όμως αυτό δεν φτάνει και αυτό ισχύει για όλους τους οργανισμούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη ΣΕΠΟΛ, έλαβε 2,5 εκατομμύρια ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του σχεδίου για την καταπολέμηση της θερμοκρατίας και για την ε, ολοκλήρωση των ε, εκπαιδευτικών δυνατοτήτων στη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Αφρική. Όμως δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για το πού πήγαν αυτά τα χρήματα πού διοχετεύτηκαν αυτά τα ποσά. Όντω συνέβαλαν στην καταπολέμηση τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι σαφέ. Το ίδιο ισχύει και για τους αξιωματούχους ε, που, ε, μάλλον που ε, εκπαίδευσε η ΣΕΠΟΛ το 2015 Χιλιάδε αξιωματικοί λοιπόν ε, πέρασαν αυτή την εκπαίδευση, αλλά δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Ε, δεν υπάρχει κάποια αξιολόγηση για να ξέρουμε κι εμείς αν όντω απέφερε αυτή η κατάρτιση κάτι. Τίποτα δεν έχουμε. Και έχουμε και μία σύσταση για όλους τους οργανισμούς. Θεωρώ ότι θα πρέπει στον ιστότοπό του να αναφέρουν την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την κάθε υπηρεσία. Οι εκθέσει αυτέ ε, βέβαια μπορεί να τι βρει κανεί ε, στον ιστότοπο του ελεγκτικού συνεδρίου. Αλλά θα πρέπει και στον ιστότοπο του εν λόγω οργανισμού να υπάρχει η σχετική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, και ένα αρνητικό σχόλιο αν θέλετε. Για παράδειγμα τώρα που συζητούμε τέτοια ζητήματα για τους οργανισμούς, δεν υπάρχει κανένας εκπρόσωπος των Ευρωπαϊκών Οργανισμών εδώ στην αίθουσα. Βλέπω μόνο κενέ θέσεις. Δεν ξέρω αν δεν τους ενδιαφέρει η επιλογή, τη θεωρούν δεδομένη, την απαλλαγή. Όπως και να έχει, δεν είναι φυσιολογικό. Ευχαριστώ. Okay, ευχαριστώ πολύ κύριε Μάκοβεϊ. Νομίζω ότι όντω ε, δεν υπάρχει κανείς εκπρόσωπος από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Α, υπάρχει ένας. I'm just trying to check which agency is present, but there is one. Uh, there is one, yeah. I think you've made your point. Ναι, υπάρχει ένας, αλλά έχετε δίκιο όντως. Για την ακρίβεια όμως να πούμε ότι υπάρχει ένας. Επομένω η Γιουλίζα είναι η μόνη που θέλει να πάρει την απαλλαγή. Ναι, νομίζω ότι ήταν εύστοχη η παρατηρήσή σας. Ευχαριστούμε και την Γιουλίζα που είναι εδώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τζέζεκ ήταν συγητής και εσείς, Τζεράρντ, ε, τον αντικαταστήσατε επάξια, αλλά δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο. Κύριε Πρόεδρε, με τα χαράς ε, θα απαντούσα σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό ο ρόλο μου. Θα μεταφέρω όμως πιστά ε, τα όσα αναφέρατε ε, στο συνάδελφό μου Πίτερ ε, Γέζεκ και επιβεβαιώνω ότι θα είναι και στη διάθεση όλων των σχεδόν εισηγητών για να συζητήσει όλες τις πιθανές τροπολογίες ως προς τις εκθέσεις του. Σας ευχαριστώ πολύ, Ζεά. που τον αντικαταστήσατε για να ακολουθήσουμε και το χρονοδιάγραμμα. Υπερθυμίζω μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, 7 το απόγευμα. Και ελπίζουμε να περάσουμε σε ψηφοφορία στις 9 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης για τη συμβολή τους σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 21. προσχέδιο σχέδιο γνωμοδότηση σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Λιχτενστάν για συμπληρωματικού κανόνε σχετικά με το μέσο χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερική Ασφάλεια για την περίοδο 2014-2020. Η συγκητή είναι ο κύριο Γιώζεφ Βάιντεν Χόλζερ. Δεν ξέρω αν ε, κάποιο τον ε, αντικαθιστά. Μπορούμε να το περάσουμε. Δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 18 Ιανουαρίου. Θα δω. Αλλά ας περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 22. Συναδελφοί, ελέγχουμε αν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο ε, σημείο για την ιδιωτικότητα ή όχι. Ένα λεπτό, δώστε μου. As I was saying, <laughs> sorry, um, colleagues thought that uh, we needed some... Uh, Ωραία. Κάποιοι θεωρούσαν ότι πρέπει να παρευρίσκονται και άλλοι συνάδελφοι για την ασπίδα προστασία για την ιδιωτικότητα, αλλά δεν χρειάζεται. Σημείο 22, λοιπόν. Επάρκεια τη προστασία που παρέχεται από την ασπίδα προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα, για την ιδιωτικότητα. Πρόκειται για σχέδιο ψηφίσματο. Μερικέ παρατηρήσει να κάνω πριν δώσουμε το λόγο στου συναδέλφου. Θα θυμάστε ότι μετά την υιοθέτηση από την Επιτροπή της Συμφωνίας ε, Επάρκειας ε, για την ε, ασπίδα προστασία Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑ. Στι 4 Ιουλίου οι συντονιστέ αποφάσισαν να, προχωρήσουν σε ένα σχέδιο ψηφίσματο. Πρόκειται λοιπόν για αποτέλεσμα δουλειά μεταξύ διαφόρων πολιτικών ομάδων. Πρόκειται για ένα ισορροπημένο κείμενο που αντικατοπτρίζει τις επιμέρους θέσεις που έχουν οι πολιτικές ομάδες. Ε, σχετίζεται και με την ε, ομάδα εργασία του άρθρου 29 και το ψήφισμα του Μαΐου του 2016 για τις πρατηλαντικές ε, ροές δεδομένων. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τις βελτιώσεις του τελικού κειμένου της ασπίδας προστασίας σε σχέση με, το προηγούμενο, με την προηγούμενη πρόταση για τον ασφαλή λιμένα ε, θεωρούμε ότι θα διευκολύνει τι ε, ανταλλαγέ δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, συγκεκριμένα από μικρέ επιχειρήσει ε, και ότι οι εποπτικές ε, αρμοδιότητες ε, δεν θα επηρεάζονται από την απόφαση επάρκειας. Ε, λαμβάνει υπόψη και τις διευκρινήσει και ερμηνείες της ε, αμερικανική κυβέρνηση και ιδίω ό,τι αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις ε, μυστικέ υπηρεσίε και τις αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία του συνηγόρου του πολίτη. Επίσης, εντοπίζονται και ζητήματα προβληματισμού που εκκρεμούν ή δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί, είτε πρόκειται για εμπορικέ πτυχές, είτε για τις και τις πτυχές που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και των αρχών επιβολής του νόμου. Αυτό αντικατοπτρίζει και τα όσα εξετάζονται από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Ε, τέλος, καλούμε την Επιτροπή να διεξαγάγει πλήρη και εμπεστατωμένη εξέταση όλων των ελλείψεων και ανεπαρκειών που εντοπίζονται με πλήρη ε, συμμετοχή ε, των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων και με πλήρη πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο και σε εγκαταστάσεις προκειμένου να γίνει σωστή αξιολόγηση και καλή και τις Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων να διασφαλίσουν ότι οι υποπτικές τους εξουσίες τηρούνται και γίνονται σεβαστές. Αυτά ήθελα να πω για το σχέδιο ψηφίσματος. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συντονιστέ ε, της ΛΥΜΠΕ και βέβαια και στα μέλη ε, για τα σχόλιά τους. Με ενημέρωσαν ότι δεν έχει έρθει ακόμα ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έρθουν όμως σύντομα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση με τους συναδέλφου γιατί είναι και πέμπτη απόγευμα και θέλουμε να τελειώνουμε όσο γίνεται νωρίτερα. Να μην σας καθυστερήσω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο κύριος Μπόνι έχει το λόγο. If you want to speak first, please. You ready? Did, did you not hear me or? Yeah. No, Mr. I think you, you see, I, I always suspected. Κύριε Μπόνη, πάντα έχω αυτή την υποψία ότι κάποια μέλη δεν με ακούν και δεν με προσέχουν και τώρα βγήκα σωστός τελικά. Μάλλον κάνατε κάτι άλλο πιο ενδιαφέρον. Είπα λοιπόν ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα φτάσει και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εφόσον ε, έχουμε εδώ μαζί μας ε, μέλη του Κοινοβουλίου, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και σας έδωσα το λόγο. Να είστε πρώτος, κύριε Μπόνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Θα πάρω το λόγο τώρα πριν φτάσει η Επιτροπή, γιατί μάλλον δεν είμαι έτοιμο να του αντιμετωπίσω. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Πρέπει να εξετάσουμε δύο πτυχές. Αφενός, χρειαζόμαστε την ε, ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα για να κάνουμε τις ε, σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένων Πολιτειών όσο γίνεται πιο ανοιχτές και διαφανείς. Συμφωνώ λοιπόν ε, σε ό,τι αφορά ορισμένες ανησυχίες και προβληματισμούς, με άλλα όμως δεν συμφωνώ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη διατύπωση. Αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα. Μπορούμε να τα συζητήσουμε, και εγώ και άλλοι θα υποβάλουμε ε, τροπολογίες και το συζητάμε μετά. Το πραγματικό πρόβλημα είναι τι θέση θα λάβει η νέα Αμερικανική κυβέρνηση έναντι αυτής της ε, ασπίδας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση πριν από μερικούς ε, μήνες κατά τη διάρκεια του IGF. Ε, και η πολιτική μαμάδα ομάδα και η εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα συζήτησε όλα αυτά με μια αποστολή των ΗΠΑ και τους ρωτήσαμε ποια είναι η γνώμη τους ό,τι αφορά την διατήρηση λύσεων που είχαμε βρει σχετικά με επιμέρους ε, ζητήματα. Και εκείνοι μας είπαν ανοιχτά ότι δεν γνωρίζουν. Γιατί θα αναλάβουν νέα πρόσωπα, για παράδειγμα στην NSA, στη CIA κτλ. Προτείνω λοιπόν να εξετάσουμε μεν το σχέδιο ψηφίσματος, αλλά να δούμε μήπως σε κάποιους τομείς να περιμένουμε να υποβάλουμε νέα ζητήματα στη νέα διοίκηση, στη νέα κυβέρνηση ή να περιμένουμε ένα δύο μήνες για να δούμε ποια θα είναι η στάση της νέας ε, διοίκησης. Υπάρχει λοιπόν ένα ερωτηματικό γιατί με αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα. Στις 20 Ιανουαρίου αναλαμβάνει η νέα κυβέρνηση της κι Ευχαριστώ αγαπητέ Βόνη. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δεν μίλησα εγώ για την νέα κυβέρνηση βέβαια στην εισαγωγική μου τοποθέτηση. Αναγνωρίζετε νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και κάποιες διαφωνίες σχετικά με το ε, ποια είναι τα βασικά θέματα μέσα στις διάφορες πολιτικές μας ομάδες ποια είναι θετικά και αρνητικά σημεία. Θα τα δούμε αυτά στη συζήτηση, αλλά λέτε και κάτι ξεχωριστό. Σημαντικό άλλωστε, σχετικά με την αλλαγή των προσώπων στην Αμερικανική διοίκηση. Βέβαια, οι συνάδελφοί μας θα υποβάλουν τροπολογίες. Και ω Επιτροπή μεταβαίνουμε στι Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο, 7ο μήνα. Και Θα ήθελα ωστόσο να ακούσουμε και τις απόψεις των συναδέλφων σήμερα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και ευχαριστώ που θέσατε το θέμα. Μπριγκίτε, εσείς νομίζω τώρα, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Πρώτα, επανέρχομαι στο 21. Ίσως μπορούμε να το πούμε, να το συζητήσουμε αργότερα, διότι αρχικά είχε ανακοινωθεί για τις 4 το απόγευμα και μπορεί ο εισηγητής ή η εισηγητρία να έρθει αργότερα. Σε ό,τι αφορά το ψήφισμα για το Privacy Shield, πρώτη ερώτηση. Γιατί να συζητήσουμε διάφορες διατυπώσεις που ενδέχεται να είναι πιο απλές ή λιγότερο απλές, όταν εν τέλει το ψήφισμα δεν πρόκειται να επιφέρει καμιά διαφορά, διότι έχει εγκριθεί η προστασία Τη ε, προσωπική σφαίρα και ό,τι και να αποφασίσουμε δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Τώρα, υπό τον τίτλο αυτό, εγώ δηλώνω σχετικά ικανοποιημένη με το κείμενο του ψηφίσματος. Και νομίζω ότι αρχίζουμε με έξι πολύ θετικά σημεία. Δέστε εκείνα τις παραγράφους εκείνες που έχουν τους αριθμούς 9-18. Ο δε αγαπητός Μπόνι θα είναι και αυτός νομίζω πολύ ευχαριστημένος. Όμως έχουμε και τέσσερα σημεία κριτικής. Είναι σημαντικά βέβαια, ιδίως για την δυνατότητα που εξακολουθεί να υφίσταται συλλογής χίδιν δεδομένων. Κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και πάλι. και κάτι που δεν έχει απόλυτα ξεκαθαριστεί της αποτελεσματικής δικαστικής επανόρθωσης και για τον Ombudsman ή Ombudswoman. Και έχουμε και ορισμένα σημεία κριτικής. Είναι περιορισμένος ο ρόλος του Κοινοβουλίου μέσα στην διαδικασία της έκδοσης των αποφάσεων και θα επανέλθουμε αργότερα, νομίζω θα επανέλθω και εγώ δηλαδή, τι έγινε με την απόφαση περί ασφαλούς λιμένος. Το επόμενο θέμα σχετικά με το τι να κάνουμε με την επανεξέταση και να έχει κάποιους στόχους που θα ελέγχει η Επιτροπή μας, όπως η απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα εγγραφά και εγκαταστάσεις και πλήρης εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα βήματα της κοινή ετήσιας επανεξέτασης. Ένα σημαντικό θέμα, ίσως είναι φοβούμε αλλά ελπίζω όχι, ελπίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα όπως με τον ασφαλή λιμένα, Safe Harbor, όπου διαπιστώσαμε σε πρώιμο στάδιο ότι δεν λειτουργούσε και το είχαμε, είχαμε τονίσει τότε κάποια πραγματικά εφιστάμενα προβλήματα ξανά και ξανά τα τονίσαμε αυτά χωρίς όμως να γίνει τίποτε και μόνο όταν ένας ιδιώτης προσέφηκε σε δικαστήριο αρχίσαμε κάποιες διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κειμένου αυτό δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί ελπίζω αυτή εδώ η ασπίδα προστασίας να λειτουργήσει καλύτερα από τον ασφαλή λιμένα διότι όπως είπα έχουμε ακόμα πηγές ανησυχίας μέσα στο κείμενο. Εάν ανακύψουν προβλήματα, το μόνο που μπορώ να πράξω είναι να ζητήσω από όλους όσοι συμμετέχουν στην επανεξέταση αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε προβλήματα ενδεχομένως να προκύψουν και να μην κρυφτούμε πίσω από τον ισχυρισμό ότι χρειαζόμαστε ανταλλαγή δεδομένων, πράγμα το οποίο αληθεύει αλλά να ψάξουμε να βρούμε λύσεις και να βάλουμε ε, και να προστατεύσουμε την προσωπική σφαίρα των πολιτών μας. Ευχαριστώ, Μπριγκίτε. Η Σοφή Ιντεφέλντ. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Ούτε ξέρω πόσες φορές έχουμε συζητήσει τις μεταφορές δεδομένων μεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού. Ήλπιζα ότι θα είχαμε επιτέλους μια ρύθμιση που θα ήταν ε, υδατοστεγής και θα επέτρεπε την ανταλλαγή δεδομένων χωρίς πρόβλημα. Φαίνεται όμως ε, ότι ε, ε, αυτό το δράμα συνεχίζεται. Όπως είπατε κι εσείς, η συζήτηση αυτή προβλεπόταν αρχικά για τις 4 και 4. Εγώ βιάστηκα και ήρθα, αλλά είμαι βεβαία ότι θα αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωση, η οποία βεβαίως δεν είναι εδώ ακόμη και με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένω τι θα πει. Έχω και κάποιε ερωτήσει. Εφόσον έρθουν, να τους ρωτήσουμε. Αν όχι, να ζητήσουμε γραπτή απάντηση. Οι, ερώτηση, ερωτήσεις μου έχουν ω εξή. και μπορούμε ίσως να, να τις εντάξουμε και ε, υπομορφή τροπολογίας στο ψήφισμα. Πρώτα λοιπόν, και πέραν από την ε, μετάβαση σε νέα Αμερικανική κυβέρνηση, η Ευρωπαία Επίτροπος, κυρία Γιάροβα, εξεδήλωσε έλλειψη ικανοποίησης από την Αμερικανική απάντηση σχετικά με την υπόθεση του Yahoo που ε, υποχρώνεται να σαρώνει τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, να κάνει σκάν στα email. Αυτό θα έχει επιπτώσεις σε θέματα προσωπικής σφαίρας. Ελπίζω να μην ακολουθήσουμε την ίδια οδό όπως με τον ασφαλή λιμένα που αποδείχθηκε η ε, οδός ε, ότι υπελείπετο δεν ήταν δηλαδή ικανοποιητική. Ελπίζω ότι θα λάβουμε περισσότερες πληροφορίες για τη νέα κυβέρνηση και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα πρόσωπα αυτής, ιδίως ό,τι αφορά την αντικατάσταση της κυρίας Νοβέλη, αυτήν την ονομαζόμενη Ombudsman, ποιες ε, εγγύησεις λαμβάνουμε για την ανεξαρτησία του Ευρωπαίου Ombudsman, και τι γίνεται με την πρόταση του υποψηφίου Προέδρου Τραμπ για τη δέσμευση ότι θα επανεξετάσει την ε, οδηγία υπαριθμών 28 της Αμερικανικής κυβέρνησης γιατί ε, βλέπουμε διάφορες προφορίες να κυκλοφορούν στον τύπο σχετικά με την νέα Αμερικανική κυβέρνηση και εκεί αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα ήθελα να γνωρίζω ακόμη λίγο περισσότερα για μια ανακοίνωση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του την εβδομάδα σχετικά με εμπορικούς εταίρους Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, χώρες όπως Ιαπωνία, Κορέα και άλλες, σχετικά με ρυθμίσεις παρόμοιες με αυτές της ε, ασπίδας προστασίας. Θα ήθελα να μάθω και για αυτά λίγα περισσότερα. Μία τελευταία ερώτηση. Είδα κάτι, αν και δεν μπόρεσα να εξετάσω τις λεπτομέρειες, ανακοίνωση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, χρήση δεσμευτικών κανόνων σε εταιρείε για την μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στις δύο του Ατλαντικού και μήπως η Κομισιόν αποφάσισε να μετακινήσει την έμφαση από την ε, ε, ασπίδα προστασίας προσωπικής σφαίρας προς δεσμευτικούς κανόνες για τις επιχειρήσεις. Τέλος, κάτι που εν μέρη ε, προσκείται σε αυτό. Η συνολική αυτή συμφωνία έχει κοινοποιηθεί, μεν δεν έχει όμως υπογραφεί, δηλαδή βρίσκεται στα ράφια για κάποιο διάστημα. Θα ήταν σωστό να λάβουμε κάποιες πληροφορίες και για το καθεστώς αυτού του φακέλου. Πρόεδρος Μωράης, ευχαριστώ. θα έπρεπε να είχαμε περιμένει. Προχωρούν τα πράγματα σύντομα. Βέβαια είναι και πέμπτη απόγευμα. Αρχίζει και αυξάνει ο ρυθμός της καρδιάς και η αδρεναλίνη. Όλα τα πράγματα πηγαίνουν γρήγορα. Όλοι σκέφτονται το ταξίδι επιστροφής. Αλλά τελικώ ήταν ίσω λάθο που αρχίσαμε τη συζήτηση χωρί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στο μεταξύ όμω έχει έλθει. και δεν θα ήταν και δίκαιο απέναντι στον κύριο Τζανκαρέλη να κληθεί να απαντήσει χωρίς να έχει ακούσει τις ερωτήσεις. Ακούσα πρώτα τον κύριο Βόσ. Και για χάρη της Επιτροπής, αν θέλετε, εσείς θα επαναλάβετε πολύ σύντομα τα βασικά που είπατε. Και μετά θα προχωρήσουμε σε άλλο γύρο, γιατί έχουμε χρόνο. Άξελ Φως. Είστε και ο τελευταίος στον κατάλογο. Ευχαριστώ. Πρώτα, ερώτημα. Θέλουμε διατλαντική μεταφορά δεδομένων ναι ή όχι. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλουμε. Διότι αναμένουμε ορθή διαχείριση των δεδομένων. Θέλουμε και εθνική ασφάλεια που απαιτεί κάθε χώρα μέλος και βέβαια και οι Ούτε και εκεί μπορεί να έχει κανείς αντίρρηση, διότι οι κίνδυνοι και οι απειλές είναι γνωστά. Άρα είναι καθήκον μας να αναζητήσουμε μια ισορροπία στον ε, τομέα αυτό. Το κάναμε αυτό και πέρσι μάλιστα. Συζητήσαμε απειράκι το θέμα αυτό. Μας απάντησε με ώρες ολόκληρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ακούσαμε αυτά τα πράγματα ξανά και ξανά. Το θέμα αυτό θεωρώ ότι το έχουμε κλείσει. Διερωτώ δηλαδή γιατί συζητούμε πάλι αυτό το ψήφισμα. Βεβαίως πάντοτε μπορεί κανείς να αλλάξει κάποιες λεπτομέρειες σε μια ισορροπία η οποία ήδη εξευρεθεί. Μπορεί να ασκήσει κάποια κριτική διότι κάποιος ή κάποιος άλλος δεν είναι ικανοποιημένοι απολύτως. Και βεβαίως και το δικαστήριο ενδέχεται να εγκύψει σε αυτήν. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε μια βάση. Και γι' αυτό άλλωστε το λόγο καταλήξαμε σε, όπως είπα, μία βάση και είπαμε ότι κάθε χρόνο θα γίνεται η εποπτεία, ο έλεγχος, η επανεξέταση και θα επιφέρονται οι αλλαγές. Και εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με έναν από τους τρόπους αυτούς. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο επανερχόμεθα σε κάτι το οποίο ήδη έχει κρυθεί. Εάν φοβούμεθα την πολιτική ευθύνη, ε, νομίζω ότι αυτό δεν τιμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί κάποια πράγματα να μην απόλυτα ε, υδατοστεγή ε, από άποψη νομική απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και χρειάζεται να λάβουμε την ευθύνη, διότι η ζωή συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δύο χρόνια μέχρι ότου να υπάρξει κάποιο είδους βάση νομικά διατυπωμένη η οποία να μας απασχολήσει ξανά. Χρειάζεται να λάβουμε και κάποια ευθύνη απέναντι στο κοινό, απέναντι στην οικονομία. Όλα αυτά προσπαθήσαμε να τα κάνουμε με τούτην εδώ την Privacy Shield και κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι εν πάση περιπτώσει δεν αποτελεί και την απολύτως τελεσίδικη λύση, πρόκειται για μια αφετηρία. αφετηρία. Και αυτή θα διαμορφωθεί ξανά και ξανά καθώς εμφανίζονται τα προβλήματα. Δεν θα συμφωνήσουμε λοιπόν με το ψήφισμα, εκτός εάν υποβληθούν κάποιες συγκεκριμένε συμβαστικές διατυπώσεις. Κατά τη γνώμη μου, εάν δεν συμβεί αυτό, το όλο εγχείρημα είναι απολύτως περιττό. Όπως είπα, χρειάζεται μια βάση και όχι να ψάχνουμε από εδώ και από εκεί. Οι Αμερικανοί έχουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες ασφαλείας να λέμε ότι ξανά και ξανά ναι, άλλο ένα βήμα και άλλο ένα βήμα και άλλο ένα βήμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε ότι ναι, πρόκειται για μια αφετηρία η οποία θα εξελιχθεί. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με την, ε, με την ε, ασπίδα προστασίας προσωπικής σφαίρας. Δεν μας αρέσει το ψήφισμα. Χρειάζεται να εξευρεθούν κάποιοι συμβασμοί. Αλλιώς δεν θα πρέπει να περιμένετε υποστήριξη εκ μέρους μας. Σας ευχαριστώ, Άξελ. Ε, καλά είναι να λέτε τα πράγματα όπως τα αισθάνεστε. Είναι διαδικαστικό, Birgit. Η γενική παρατήρηση. Χωρίς μικρόφωνο η Birgit δεν ακούγεται. Μίλησες πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε είναι δίκαιο αυτό που ζητάς και όσοι συνάδελφοι πήραν το λόγο μπορούν να τα ξαναπούν εφόσον το κάνουν με συνοπτικό τρόπο. Κύριε Ζήπελ, θα ήθελα να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι υπάρχουν πολλά θετικά στο ψήφισμα αυτό και δεν καταλαβαίνω γιατί ε, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε και από τις άλλες πολιτικές ομάδες ότι υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες και κάποια θέματα ανοιχτά. Δεύτερον, δεν δέχομαι εγώ την ε, παρατήρηση ότι κάνουμε κριτική μόνο και μόνο γιατί αυτό είναι μια συμφωνία ανάμεσα στην Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Αυτό είναι απαράδεκτο, δεν μπορούμε να το δεχτούμε και δεν θα πρέπει να ακούγονται τέτοια πράγματα. Επανερχόμενος τώρα στην ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να μάθω συγκεκριμένα αν θα μπορούσε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στα πλαίσια της συνεργασίας για την επανεξέταση της ασπίδας αυτής της προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων και στο πλαίσιο της συνεργασίας Επιτροπής και Κοινοβούλια. Έχετε κάποιο σχέδιο, κάποια διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε με διαφορετικό τρόπο όταν ξεκινήσουν διαφορετικού τύπου ανησυχίες. με διαφορετικό από ότι, τρόπο από ό,τι έχει συμβεί στους ασφαλείς λιμένες. Η κριτική μας δεν λήφθη σοβαρά υπόψη και τώρα το πληρώνουμε. Λοιπόν, ε, πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανησυχίες αυτές διασφαλίζοντας τη σωστή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Τα υπόλοιπα μέλη, αν θέλουν συμπερασματικά να θέσουν τα θέματά τους στην Επιτροπή, ζητώ συγγνώμη για τη διαδικασία. Δεν ζητά κάποιος το λόγο. Σοφή, θες να επαναλάβεις ίσως αυτά τα οποία είπες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνθετικά παρακαλώ. Μπορώ να του στείλω ένα mail λέει η Σοφή. Καλώς, όπως θέλετε. Αν περάσω τώρα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπαθώ να είμαι δίκαιος και μπερδεύομαι. Δεν θέλω να χειροτερεύσω τις συνθήκες συζήτησης, να πω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το αν θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν σίγουρα πολλά θετικά στην πρόταση. Αλλά θα υπάρξουν και πολλαπλές αναθεωρήσεις στο μέλλον. Και γι' αυτό καλό είναι να έχουμε ένα έγγραφο το οποίο να αποτυπώνει την τρέχουσα εικόνα της θέσης του Κοινοβουλίου σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος να γίνει κάτι τέτοιο και μετά από τις τροπολογίες θα πρέπει να δούμε ακριβώς πού θα ισορροπήσει η ζυγαριά. Γι' αυτό δίνω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μας πει την άποψή της. Ευχαριστώ. Έφτασα με καθυστέρηση κι εγώ. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις που άκουσα. Ε, ίσως να μην είμαι πλήρης στις απαντήσεις ε, και ε, μπορείτε να τις θέσετε εκ νέου τις ερωτήσεις σας. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με την μελλοντική διαχείριση ή μάλλον με τη μελλοντική Αμερικανική κυβέρνηση και τι επιπτώσεις θα έχει η καινούργια κυβέρνηση στα θέματα της ασπίδας. Εδώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να μεταφέρω τις απόψεις μου σε κάποια θέματα. Να μην ξεχνάμε ε, το τι είναι η ασπίδα αυτή προστασίας. Βασίζεται σε υποχρεώσεις ανηλυμένες και δεσμευτικές για τη ΣΥΠΑ. Όχι την μία κυβέρνηση ή την άλλη. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια που έγινε είναι να καταλήξουμε σε ένα ωφέλιμο και για τις δύο πλευρές θέμα ε, φυσικά τίθεται το θέμα της συζήτησης, της συνέχισης των υποχρεώσεων αυτών. Αλλά αυτό άλλωστε αποτελεί και ένα κίνητρο έτσι ώστε να σεβαστούμε τις αποφάσεις που έχουμε λάβει. Να πω επίσης ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι υποχρεώσεις αυτές δεν τηρηθούν, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι πλέον κανόνες στην διάθεσή μας που διευκρινίζουν ακριβώς το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε και ε, τι μπορούμε να πάρουμε σαν μέτρα τα οποία ακριβώς να ανταποδίδουν αν θέλετε τη μη τήρηση των συμπεφωνημένων. Αυτή είναι θα έλεγα η βασική δομή και οι κανόνες πάνω στους οποίους βασιζόμαστε και με την προηγούμενη κυβέρνηση στη ΣΥΠΑ και με τις επόμενες όποιες και αν είναι αυτές. Να πω επίσης ότι το να προσπαθήσουμε να θεωρήσουμε σταθερά τα θεμέλια αυτής της ασπίδας προστασίας δεν είναι μόνο ένα σαφές μήνυμα το οποίο έχουμε στείλει στην κυβέρνηση του, ε, των ΗΠΑ, αλλά και στα μέλη του Κογκρέσου. Είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο και σαφές στους Αμερικανούς συνομιλητές μας. Ένα μικρό παράδειγμα. Ο βουλευτής της Βουλής των Αντιπροσώπων έστειλε μία επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ όχι μόνο να υπογραμμίσει τη σημασία του Privacy Shield, αλλά υπογράμμισε στην επιστολή αυτή ότι πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται, να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εποπτείας και του ελέγχου που βρίσκονται στη βάση της ασπίδας προστασίας των ιδιωτικών στοιχείων και δεδομένων γιατί αλλιώς δεν θα επιβιώσει η ασπίδα αυτή. Αυτό θα έλεγα δείχνει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν ε, βελτιώσει την κατάσταση, έχουν εδρεωθεί πλέον ε, ε και νομίζω ότι θα πρέπει να αγκυρωθούμε ακόμα περισσότερο σε αυτές γιατί θα πρέπει να καταλάβουν στο Κογκρέσο ότι αν ένα βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αυτής εγκαταλειφθεί, αυτό θα έχει πραγματικά πολύ συγκεκριμένα αρνητικά αποτελέσματα για το θέμα της ασπίδας. Κατά τα άλλα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει η καινούργια κυβέρνηση, έχουμε όμως συγκεκριμένες συμφωνίες, μηχανισμούς που θα μας επιτρέψουν να αντιδράσουμε στην περίπτωση κατά την οποία κάτι αλλάξει μονομερός. για την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται από τη Συμφωνία ότι στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης θα προετοιμάζει μία έκθεση η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μετά την αναθεώρηση, πριν. Θα συνεχίσουμε τον διάλογο τον οποίο έχουμε, ακόμα και σήμερα αυτό κάνουμε. Θα σας ενημερώσω και πριν το τέλος του μήνα. Και θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε και τις απόψεις του Κοινοβουλίου για τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Να σας διαβεβαιώσω πάντως ότι η εποπτεία της εξέλιξης της διαδικασίας και το θέμα της συνεχιζόμενης τήρησης των συμπεφωνημένων είναι κάτι το οποίο δεν θα μας απασχολήσει μόνο στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης, αλλά με συνεχή τρόπο. Υπήρξαν επίσης, αν κατάλαβα καλά, αναφορές και στην ανακοίνωση του συνόλου των επιτρόπων πριν δύο μέρες και που ε, αναφέρονται σε αντιστοιχήσεις επάρκειας με χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Αυτό αντικατοπτρίζει ότι η Ιαπωνία και η Κορέα πρόσφατα εξυγχρόνισαν τους νόμους ε, περί ιδιωτικότητας και υιοθέτησαν νόμους και νομίζω ότι οι νόμοι αυτοί συγκλίνουν και αποτελούν στοιχεία ενοποίησης και κοινά στοιχεία με τις δικές μας νομικές ρυθμίσεις. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ε, ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τη σύγκληση αυτή και να πάρουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις για την αναγνώριση της επάρκειας των μέτρων των χωρών αυτών. Πάντως είμαι στη διάθεσή σας πάντα για να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις που πιθανώς παρέλειψα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις σε σχόλια. Στον κύριο Καρέλη, ο κύριος Βάντερ Χόλουζερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όχι, δεν περνάμε στο επόμενο. Απλώ ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν ε, άλλα σχόλια για τον κύριο Καρέλη. Εάν όχι, να επισημάνω ότι ανέφερε και ο ίδιος ότι η κυρία Γιούροβα θα έρθει ε, στις 23 Ιανουαρίου και θα ήθελα να αναφέρω ότι μέχρι τι 19 έχετε προθεσμή υποβολή στραβολογιών. Καλό θα ήταν να την μεταθέσουμε για τις 24 λοιπόν. Να ακούσουμε πρώτα λοιπόν να συζητήσουμε την κυρία Γιούροβα και μετά να το ξαναδούμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσεί. Να πάει λοιπόν η προθεσμία για τις 24. Ωραία. Και εγώ Είπα πριν ότι το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε αναθεωρήσεις και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καρέλη πότε θα γίνει η, η επόμενη αναθεώρηση. Φέτος, αν κατάλαβα καλά. so it will take place. Ναι, φέτος βέβαια. Το σημαντικό είναι, όπως ξέρετε, ε, πρέπει πρώτα να διοριστούν και οι συνομιλητές μας από αμερικανικής πλευράς, αλλά θεωρούμε ότι θα φτάσουμε τον Αύγουστο, εκεί κλείνει το ο χρόνος λοιπόν, μάλλον το Σεπτέμβριο λοιπόν θα γίνει η αναθεώρηση και έτσι θα έχουμε το χρόνο για να οριστούν τα νέα πρόσωπα στην Αμερικανική κυβέρνηση και να έχουμε να αποκτήσουμε και κάποια εμπειρία μέχρι το καλοκαίρι για την υλοποίηση. Ε, και έτσι μετά να έχουμε την αναθεώρηση. Κάτι τελευταίο από την κυρία Εντφέλτ. Προηγουμένως μίλησα για την ε, συμφωνία Ομπρέλα και εφόσον είστε και εδώ, επί τη ευκαιρία μπορείτε να μας ενημερώσετε για αυτό το ζήτημα, γιατί παρότι δεν είμαι νομικός, κατανοώ ότι η κύρωση έχει γίνει ήδη, αλλά και πάλι θα πρέπει να υπάρξει κοινοποίηση και αυτό δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω πώς ε, ακριβώς πάει. Και αν αυτό γίνει πριν ε, καταφτάσει η ε, νέα κυβέρνηση Τραμπ ή όχι. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε λοιπόν. Παρακαλώ. Μάλιστα, με τα χαράς. Να σας πω δύο λόγια γι' αυτό. Δεν είστε νομικός, αλλά είναι νομικό το ερώτημα. Γι' αυτό και ως νομικός ε, θα απαντήσω και πολύ συγκεκριμένα. Η εσωτερική διαδικασία για την ε, ε ολοκλήρωση της ε, ομπρέλας έχει γίνει και από τις δύο πλευρές. Η δική σας ψήφος λοιπόν για την Ευρώπη και η απόφαση του Συμβουλίου. Έχουμε αρχικά τη σύναψη τη συμφωνία λοιπόν, μετά όμω είναι άλλο η θέση σε ισχύ. Για να τεθεί σε ισχύ η Ομπρέλα λοιπόν, χρειαζόμαστε, όπω ξέρετε πολύ καλά, τις απαραίτη, τους απαραίτητους που πρέπει να γίνουν από την Αμερικανική κυβέρνηση ε, για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας ε, θα υποφελούνται από, την, τον νόμο ε, δικαστικής προσφυγής και τον νόμο μονοδών. Θέλουμε λοιπόν να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία μόνο όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το βήμα του ορισμού. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι οι συνομιλητές μας, ιδίως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ε, προβαίνει σε αυτούς τους διορισμούς. Στην τελευταία διπουργική ε, διάσκεψη το Δεκέμβριο ε, η Γενική Εισαγγελέα, κυρία Λίντς, είπε ότι επεδίωκε να ολοκληρωθούν αυτοί οι διορισμοί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και κατανοείτε κι εσείς και συμφωνείτε φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να γίνει σωστά και πρώτα να διοριστούν τα κατάλληλα πρόσωπα και μετά να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, 24 Ιανουαρίου είναι τελική προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Επιστρέφω στο σημείο 21, το οποίο είχε τεθεί αρχικά στις 4. Να δώσω συγγνώμη από τον κύριο Βάντερ Χόλσερ. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λίχτενστάιν για το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και το Ταμείο ασφάλειες. Ασφάλειας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόκειται για την συμμετοχή του πριγκιπάτου του Λίχτενστάιν στο Διεθνές Security Fund για το 2014-2020. Κατά βάση πρόκειται για το εξής. Το Λίχτενστάιν ως συνδεδεμένο μέλος του χώρου Σέγγεν συμμετέχει στη συμφωνία αυτή. Το Πριγκιπάτο, η Δουκάτο μάλλον, θα δει να αυξάνεται έτσι η ασφάλειά του, να ενισχύεται η ασφάλειά του για να μπορεί να εντάξει εκεί και τη διαδικασία έκδοσης προξενικών θεωρήσεων. Εν προκειμένου το Λίχτενστάιν επιθυμεί να ε, καταβάλει περίπου 200.000 ευρώ τον χρόνο στο ταμείο αυτό και πρόκειται τώρα για την χορήγηση της εγκρίσεως στην διαδικασία αυτή. Υπάρχουν δύο παράγραφοι. Η πρώτη παράγραφος λέει ότι συμφωνούμε με την ε, ε, εγκρίνουμε τη συμφωνία αυτή και η δεύτερη παράγραφος λέει ότι το, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου κοινοποιεί το κείμενο στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πριγκιπάντο του Στάιν. Άρα δεν προκύπτουν προβλήματα εδώ και νομίζω ότι δηλαδή η σύστασή μου είναι να το εγκρίνουμε το δυνατόν συντομότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών 18 Ιανουαρίου. Κοιτάζω και το ρολόι. 23, θέμα 23, το οποίο κανονικά προβλεπόταν για τις 5, μήπως μπορούμε να συμφωνείτε να το συζητήσουμε τώρα. Ο κ. Σόγκορ είναι παρόν. Δέχεστε. Πρόκειται για σχέδιο γνωμοδοτήσεως για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τουρκία για νέα συμφωνία για την επέκταση των διμερών εμπορικών σχέσεων και της Τελωνιακής Ενώσεως οι συντονιστές, οι συντονιστές της ΛΥΜΠΕ αποφάσισαν να συνταχθεί η γνωμοδότηση μόνο στα αγγλικά έργο το οποίο έλαβε ο κ. Σόγκορ που είναι και εισηγητής επομένως και παρακαλείτε να κάνει την παρουσίαση του κειμένου του. Έχετε το λόγο κύριε Σόγκορ. Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε. Αυτό είχε συζητηθεί ήδη στη διάσκεψη κορυφής της 29ης Νοεμβρίου του 2015 μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας όπου και οι δύο πλευρές δήλωσαν προθυμία να συνεχίσουν Το 2014 η, παγκόσμια, η έκθεση Παγκόσμια Τράπεζας τόνισε τα εξή θέματα. Το γεγονός ότι ορισμένοι σημαντικοί οικονομικοί κλάδοι παραμένουν εκτός οικονομική τομή εκτός Τελωνιακή Ενώσεω όπως δημόσιες προμήθειε και ενέργεια και ότι υπάρχουν ασυμμετρίες στην σχέση που οδηγεί στο ότι οι αποφάσεις για την Τελωνιακή Ένωση και σχέσεις με τρίτες χώρες αντιμετωπίζουν τις χέρι. Τα ενδεχόμενα ωφελήματα και για τις δύο πλευρές από την παράταση της Ελληνικής Ενώσεως θα ήταν σημαντικά. Εκτός από το γεγονός ότι τονίζει αυτό, η έκθεση αναφέρεται και στις προξενικές θεωρίες, θεωρήσεις, διότι η εξυγχρονισμένη ε, τελωνιακή συμφωνία θα επηρεάσει και τις εμπορικές σχέσεις, ε, της ε, μεταφορές και άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Στη βάση της τρίτης εκθέσεως προόδου και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, Υπάρχουν ακόμα 7 από τα 72 κριτήρια όπου η Τουρκία δεν έχει ανταποκριθεί για την απελευθέρωση των ξενικών θεωρήσεων και δεν θα πρέπει να ε, ε, χαλαρώσει η προσπάθεια αυτή για πολιτικούς λόγους. Ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γνωρίζουμε όλη την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ιδίω σε ζητήματα ελευθερίας έκφρασης, ε, του συνεταιρίζεστε, του συνέρχεστε και ε, ορισμένες ελευθερίες μειονοτήτων. Αν και η Τελωνιακή Ένωση δεν έχει ως άμεσο αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα και μπορεί να ισχυθεί κανεί ότι δεν έχει άμεση επίπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Πάντως εντοπίζονται σε ορισμένα ε, σημεία ε, θετικές επιπτώσεις από την Τελωνιακή Ένωση, όπως για την υγεία, για τις επαγγελματικές σχέσεις κλπ την περίπτωση μιας ενισχυμένη Ελληνική Ένωση, τα αποτελέσματα στις, στα ανθρώπινα δικαιώματα θα βελτιωθούν και από την οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό και ανεξάρτητα τώρα από την νομοδότηση της Επιτροπής ΑΦΕΤ στον τομέα αυτό και για να γίνει πιο ασφαλής η Ευρώπη και να ενισχυθεί η σταθερότητα στις γειτονικέ μας σχέσεις, νομίζω ότι είναι σημαντικό να εγκρίνουμε την νομοδοτησία αυτή και το στοιχείο των ανθρώπινων δικαιωμάτων βέβαια είναι σημαντικό για μια νέα συμφωνία. Γι' αυτό θα υποβάλω εγώ και τροπολογία προς την κατεύθυνση αυτή. Μετά από μια ενδιαφέρουσα πρώτη συζήτηση με τους κοιόδης συζητητές αναμένω τα σχόλιά σας και τη συνεργασία σας. Uh, uh, Όντως είναι σημαντικό το θέμα, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ όσοι επιθυμείτε να λάβετε το λόγο και όσοι με ακούνε βέβαια γιατί μιλώ πολύ χαμηλόφωνα. Ντόλτον, εσείς παρακαλώ πρώτος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει και ήδη μάλιστα έχει οργανώσει και σχετική συνεδρίαση μαζί μας. Από τη δική μας πλευρά νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε το σύνολο του κειμένου, το οποίο βρίσκω ότι είναι ισορροπημένο και παρόλο που θεωρώ ότι περιλαμβάνει κυρίως θέματα εμπορικών σχέσεων, που καλύτερα να τα αναλάβει η Επιτροπή ΙΝΤΑ, αλλά πάντως προσωπικά συμφωνώ με το περιεχόμενο που έχετε περιλάβει και όσα έχετε βάλει στην γνωμοδότηση. Από τη σκοπιά της ΛΥΜΠΕ νομίζω το σημαντικό είναι το ταξίδι χωρίς προξενική θεώρηση. Και αυτό εκεί πρέπει ε, να παραμείνει σταθερή στις θέσεις της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δίνεται η ελευθερία προξενικές θεωρήσεις μόνο στις χώρες εκείνες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια. Κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Τουρκίας. Μόνο 7 από τα 72 έχει εκπληρώσει η Τουρκία και είναι σημαντικό να δεχθεί αυτό και στο κείμενο. Το όλο θέμα της απελευθέρωσης των προξενικών θεωρήσεων Καλύτερα πάντω να τεθεί μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται ούτω ή άλλω μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Τουρκία. και όχι μέσα στα πλαίσια μια εμπορική συμφωνία. Γι' αυτό και ίσως ε, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να καταθέσουμε τροπολογία με σχετικό περιεχόμενο. Πέραν αυτού όμω, μα ικανοποιεί η εργασία που έχετε κάνει και όλα τα υπόλοιπα τη εκθέσεώ σα τα υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Ντάλτον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όλες τις λεπτομέρειες και εξηγήσεις που μας έδωσε αυτό το φάκελο. Εκτιμώ ιδιαίτερως και την ε, μνήα που έκανε ε, στην πολιτική θεωρήσεων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην έκθεσή του. Επίσης, ε, ανέφερε ότι η έννοια αυτής της ανανέωσης της Θελωνιακής Ένωσης ε, επανέρχεται σε μία σύνοδο κορυφής του 2015. Και γιατί το λέω, γιατί όλοι βλέπουμε από το 2015 μέχρι σήμερα υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην Τουρκία. Και όχι προς το καλύτερο. Βέβαια, σε αυτό το κείμενο δεν μπορούμε να εξετάσουμε όλες τις λεπτομέρειες των θεωρήσεων, όμως έχω την εντύπωση ότι σε ό,τι αφορά ε, την ε, απαλλαγή θεωρήσεων για τα ταξίδια, αυτό δεν είναι ε, εξαιρετικά σημαντικό για τον Τούρκο πρόεδρο. Διαμαρτύρεται βέβαια που δεν του το έχουμε δώσει, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό για εκείνον. Πέραν λοιπόν των λεπτομεριών της Ελληνικής Ένωσης, εγώ εστιάζω την προσοχή μου στα στατηγικά ζητήματα. Θα πρέπει όντως τόσο βεβαιασμένα ε, να προχωρήσουμε αυτή την έκθεση και τη δικασία και να δώσουμε οικονομικά προνόμια σε μια κυβέρνηση που δεν σέβεται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και διαμορφώνει μια κατάσταση όπου ενδέχεται όπου όλο είναι και περισσότεροι πολίτες υπήκοοι αυτής της χώρας θέλουν να φύγουν από αυτή τη χώρα λόγω τη κατάσταση. Μήπω λοιπόν να έχουμε μια πολιτική στρατηγική να επαναφέρουμε την Τουρκία στο σωστό δρόμο. Εγώ θα πρότεινα να μην βιαστούμε, ε, να δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω σε αυτό το φάκελο, γιατί νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει πολύ περισσότερο την τουρκική κυβέρνηση παρά ε, την απελευθέρωση θεωρήσεων για τα ταξίδια. Ευχαριστώ, Μπριγκίτ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να θέλουν να πάρουν το λόγο, να δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο Σόγκουρ. Είναι μια γνωμοδότηση και τόσο λεπτό αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω κύριε Σόκουρα αν θέλετε να απαντήσετε. Δεν είστε υποχρεωμένος βέβαια. Thank you. We discussed... Ευχαριστώ. Τα συζητήσαμε ήδη και στην πρώτη συνεδρίαση. Μία πρόταση μόνο προς ε, τη συνάδελφο των σοσιαλιστών. Πράγματι, από το 2015 τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί κατά πολύ. Όμως το θέμα το θεωρήσω, νομίζω ότι όπως και να έχει, η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει τους μικρούς επιχειρηματίες. Γιατί οι μεγάλοι εντός αγωγικών έτσι κι αλλιώς παίρνουν τη θεώρηση για την Ευρώπη. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν είναι κακό να βοηθήσουμε αυτούς που Ενδεχομένω να μην ε, συμβάλλουν τόσο πολύ από πλευρά οικονομική κλίμακα, αλλά και πάλι έχουν τη σημασία του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σόγκουρ. Σίγουρα και στι συναντήσει των σκιονδών όλα αυτά θα τα συζητήσετε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 20 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα. 9 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Συνάδελφοι, τώρα για το επόμενο σημαντικό σημείο, για το άσυλο, τα σημεία 24 και 26. Είμαστε σε επαφή με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν εξελίξεις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 Sorry, this was not news about the next item. It was... Α, συγγνώμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει για το προηγούμενο ζήτημα. Κύριε Σόγκουρ, περιμένετε λίγο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσετε την απάντησή της. Α, δεν το κατάλαβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εν συντομία, λοιπόν, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ για το ζήτημα της Τουρκίας και του εξυγχρονισμού της Τελωνικής Ένωσης. Είμαι από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ήθελα αρχικά να επενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Δεκεμβρίου του 2016 υιοθέτησε την πρότασή της για σχέδιο εντολής για την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Σύντομα θα αρχίσει η εξέταση ε, της πρότασης και στο Συμβούλιο με τα κάτι και βεβαίως ε, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και την ε, εκπόνηση της ε, νομοδότησης ιδίας πρωτοβουλία από την Επιτροπή ΙΝΤΑ. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Άκουσα ένα μέρος ε, των παρεμβάσεων όταν έφτασα που αφορούσαν κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα και εγώ να επισημάνω ότι και αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι μία από τις ε, βασικές αρχές και βασικούς στόχους ε, αυτής της διαπραγμάτευσης. Ακριβώς δηλαδή η τήρηση, ο σεβασμός προς ε, τις θεμελιώδεις ε, ελευθερίες, ανθρωπινά δικαιώματα, κράτο δικαίου. Γι' αυτό προβλέπεται και στην εντολή. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο το οποίο θεωρούμε σημαντικό σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα αφορά την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας να προσθέσει και ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο ειδικά για την βιώσιμη ανάπτυξη που θα καλύπτει τέτοιες πτυχές. Σημαντικό τμήμα των διαπραγματεύσεων κατά τη γνώμη μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις και τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα να επισημάνω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικά εγχειρήματα. Βέβαια έχουμε την διαδικασία απελευθέρωσης ε, θεωρήσεων αφενός και στις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις βεβαίως ε, δεν ε, θίγουμε ζητήματα θεωρήσεων. Δεν διαπραγματευόμαστε επί τούτου. Είχαμε την πρόθεση να διαπραγματευτούμε την απελευθέρωση υπηρεσιών, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στι εμπορικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Όμω αυτό θα γίνει ξεχωριστά από τη διαδικασία απελευθέρωση θεωρήσεων. Όπω συμβαίνει με όλε τι τρίτε χώρε. Πρόσφατα παραδείγματα Βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία απελευθέρωση θεωρήσεων με τέρου όπως η Ουκρανία, η Γεωργία, με τη Μολδαβία στο παρελθόν και αυτό γινόταν ξεχωριστά από τις ε, διαπραγματεύσει για τις ε, ολοκληρωμένες εμπορικές συμφωνίες σε αυτές τις τρίτες χώρες. Επομένω, η πρόθεσή μα είναι να συνεχίσουμε να εξετάζουμε ξεχωριστά αυτά τα ζητήματα, όπω είναι παραδοσιακά η ε, τακτική μας. Ήθελα μόνο να το υπογραμμίσω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. αδελφή, για τα σημεία 24 και 26... τις παρουσιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 5 παρα 10 μου λένε ότι θα φτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανονικά πρέπει το είχαμε θέση για τις 5.30. Κάποιοι λένε ότι καλό θα ήταν να το αναβάλουμε, αλλά είναι αδύνατον. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει τέτοιος φόρτος εργασίας που δεν μπορούμε να καθυστερούμε περαιτέρω. Ήρθαμε σε επαφή λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 5 παρα 10 είναι το νωρίτερο που μπορούν να φτάσουν. Α κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα 20 λεπτών και να επανέλθουμε στι 5 παρα 10 για να δούμε αυτά τα τρία σημεία. My apologies, um, for all the... Και συγγνώμη για αυτές τις ε, αλλαγές ε, στο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το ζήτημα. 5 παρα 10 και πάλι εδώ λοιπόν.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 Καθίστε λοιπόν, συνάδελφοι, να εξηγήσω και τη διαδικασία. Και πάλι ζητώ συγγνώμη για την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα. Και γενικότερα το ότι θέσαμε για την Πέμπτη το απόγευμα και μάλιστα στο τέλος αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα. Απλώ είναι λόγω φόρτο εργασία. Θα το δείτε ότι και τη μεθεπόμενη εβδομάδα είναι πραγματικά πολύ φορτωμένη η μέσα διάταξη και γι' αυτό έπρεπε να το εξετάσουμε τώρα αυτό το σημείο κατεπηγόντω. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας λοιπόν. Θα εξετάσουμε τώρα τα σημεία 24-26. Ο κύριος Βέρβη καταφθάνει, ο κύριος Ράιαν θα μιλήσει για την μετακατάσταση, την επανεγκατάσταση και το Δουβλίνο πρώτα, αν συμφωνούν και τα μέλη. Εν είδη εισαγωγής, να πω, θα θυμάστε ότι οι τελευταίε συζητήσει ήταν με τους εκπροσώπους ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση των αποφάσεων για την μετακατάσταση και την επανακατάσταση, την υλοποίηση τη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και της ε, επανεκκίνησης ε, επιστροφών μεταναστών προ την Ελλάδα υπό το Δουβλίνο. Σε αυτή την περίπτωση η ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντική. Αρχικά επειδή η Κομισιόν προτείνει βαθμιδών να ξεκινήσουν και πάλι αυτές οι μεταφορές ε, ε, υπό το Δουβλίνο από τις 15 Μαρτίου και μετά που είχαν σταματήσει το 2011 κατόπιν δύο δικαστικών αποφάσεων ε, του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα επιστροφής μεταναστών προ την Ελλάδα, συνδέεται και με την μετακατάσταση σε αλλε χωρες χώρε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς έχουμε και το τέταρτο ε, παρά, παράρτημα μάλλον προς την τέταρτη έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Όλα αυτά εντάσσονται ε, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής ε, πολιτικής που ισχύει και για την Ελλάδα. Είναι το πιο σημαντικό θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Ιταλία το τελευταίο τρίμηνο του 2016 είχε τον υψηλότερο αριθμό αφήξεων 170.000 άτομα κατέφτασαν στο τελευταίο τρίμηνο. Μας ε, προβληματίζει ιδιαίτερως η κατάσταση στην ε, Ιταλία και πρέπει να στηρίξουμε και την Ιταλία, θεωρώ. Πρέπει να ακούσουμε και για την ανθρωπιστική κατάσταση ε, στην Ελλάδα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν αναφέρει και συνάδελφοι και μας προβληματίζει ιδιαίτερως. Και ξέρω ότι και ο κύριος Βέρβεϊ θα θέλει ε, να θίξει αυτό το εξαιρετικά ανησυχητικό ζήτημα. Και πάλι αλλάξαμε λίγο τη σειρά ε, και χαίρομαι που και οι δύο συγκεκριτές είναι εδώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. να τα κάνουμε τα πράγματα σωστά λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βέρβιν να μας παρουσιάσει την κατάσταση στην Ελλάδα και την Τουρκία για 10 λεπτά. Μετά θα περάσουμε στον κύριο Ράιεν που θα μας επισημάνει τους λόγους τους οποίους εκείνη και πάλι τη διαδικασία επιστροφής μεταναστών προς την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και τους δυο για την παρουσία σας εδώ. Ξεκινούμε με τον κύριο Βέρβη. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να καλησπερίσω τα μέλη της Επιτροπής σας, λέει ο κύριος Βέβαιη. Στις 8 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τέταρτη έκθεσή της για την Τουρκία. Επιβεβαιώθηκε η συνέχιση της παραγωγής ε, θετικών αποτελεσμάτων αλλά με πάρα πολλές δυσκολίες. Βέβαια οι μεταναστευτικές ροές ελέγχονται, είναι χαμηλές και λιγότερα είναι τα θύματα τα οποία παλαιότερα ήταν πάρα πολλά στο Αιγαίο. Υπάρχουν όμως δυσκολίες και πρέπει η συμφωνία αυτή να λειτουργήσει σε μια πιο σταθερή βάση οι σορευτικές επιπτώσεις της εφαρμογής αυτής της δήλωσης Ένωσης Τουρκίας μετά από εννέα μήνες είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Πριν εφαρμοστεί η δήλωση αυτή, πριν εννέα μήνες, After, uh, was ο αριθμός ήταν πάρα πολύ υψηλός. Τώρα πλέον μετά την εφαρμογή της συμφωνίας ο αριθμός δεν έχει ξεπεράσει τους 25 περίπου χιλιάδες. Ο αριθμός των νεκρών έπεσε από 789 σε 68 και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μείωση κατά 700 περίπου. Από 900 σχεδόν χιλιάδες λοιπόν σε 25. Βέβαια για την Ιταλία θα πρέπει να υπογραμμίσω και το έχω ήδη κάνει ότι δεν υπάρχουν πραγματικά δείγματα θα έλεγα αλλαγής της ροής εκτός από τις δεδομένες ροές στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει υπάρξει σε ορισμένους τομείς λοιπόν επιπτώσεις έχουν κατατεθεί πάνω από 11.000 αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Ε, έχουν ληφθεί ήδη 8.200 αποφάσεις σε πρώτο επίπεδο με την υποστήριξη της ΆΣΑ και 2.500 περίπου χιλιάδες έχουν εφεσιβάλει την απόφαση αυτή και σε λίγες τέτοιες περιπτώσεις έχει ήδη εκδοθεί και η απόφαση επί της εφέσεως. Για τις ε, επαναπροωθήσεις προς την Τουρκία συνεχίζονται, αλλά συνεχίζονται με έναν ρυθμό ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός. Από την 21 Μαρτίου μέχρι τώρα έχουν επιστρέψει 1247. Πολύ χαμηλότερος ο αριθμός αυτός από τις αφήξεις, παρότι οι αφήξεις είναι λιγότερες. Έχουν δημιουργηθεί αρκετά αδιέξοδα, προβλήματα σοβαρά. Να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω δύο πιο συγκεκριμένα. Πρώτον, η περιορισμένη ικανότητα εξέτασης των εφέσεων. Μια διοικητική αδυναμία εκεί, Κάναμε λοιπόν κάποια βήματα για την εξέταση των αιτήσεων σε πρώτο επίπεδο, σε πρώτη φάση, σε πρωτοβάθμιο αν θέλετε, αλλά στο δεύτερο έχουμε πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε και το οποίο εξηγεί τον μικρό αριθμό των επιστροφών είναι ότι οι δυνατότητες διοικητικές για τη λήψη των αποφάσεων για τις επαναπροωθήσεις επί των νησιών είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή διευκρινιστεί ότι ένα πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα σε άσυλο να ε, ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία και να αποφασιστεί η επιστροφή του στην Τουρκία. Το χαμηλό αυτό ποσοστό λοιπόν επιστροφών έχει αυξήσει τις πιέσεις σε ήδη ε, οριακές δυνατότητες υποδοχής στα νησιά. Οι μετανάστες αλλά και οι τοπικοί πληθυσμοί δυσφορούν όλο και περισσότερο. Αυξάνονται εντάσεις και από τις δύο πλευρές. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ίδια τη διαδικασία εξέτασης της χορήγησης ασύλου γιατί επανειλημμένα δημιουργήθηκαν προβλήματα ασφάλειας που διέκοψαν τις διαδικασίες και δημιούργησαν περαιτέρω καθυστερήσεις και περαιτέρω δυστημία. The uh, uh, είναι σαφές ότι κάποιες από τις συνθήκες uh, δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές και ιδιαίτερα είδαμε τις τελευταίες μέρες τις συνέπειες του πολύ κακού uh, καιρού που δημιούργησε σημαντικά προβλήματα. Και υπάρχει λοιπόν και αύξηση της uh, δυσφορίας του τοπικού πληθυσμού. Είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθεί κανείς με αυτά τα θέματα, γιατί είναι προφανές ότι η συνεργασία με τους τοπικούς πληθυσμούς είναι κάτι το πολύ σημαντικό και δυστυχώς καθίστανται πολύ λιγότερο δεκτικοί από ό,τι στο παρελθόν. Ο πρόεδρος σας είπε στην εισαγωγή του ότι οι εξαιρετικά κακές καιρικές συνθήκες δημιούργησαν προβλήματα και θα μου επιτρέψετε σε λίγο να σας δώσω κάποια περαιτέρω στοιχεία ενημέρωσης. Όλα αυτά λοιπόν τι δείχνουν. Απαιτούνται συμπληρωματικές προσπάθειες έτσι ώστε η παρέμβασή μας να καταστεί πιο αποτελεσματική. Και γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα νέο πρόγραμμα δράσης. Πήραμε προτάσεις και συνεισφορές από όλους τους εμπλεκομένους και οι βασικές μας δράσεις περιλαμβάνουν αυξημένους πόρους στα νησιά, αυξημένες διοικητικές δυνατότητες για τις εφέσεις, αυξημένες συνθήκες ασφαλείας, διασφάλιση αποτελεσματικών διαδικασιών επιστροφής για τους μετανάστες που δεν έχουν πλέον δικαίωμα σε άσυλο, και επίσης βελτίωση των συνθήκων υποδοχής, όπως επίσης και επιτάχυνση της επανεγκατάστασης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν, να απορροφήσουμε την καθυστέρηση που σωρεύτηκε τους τελευταίους μήνες, θέλουμε να μειώσουμε πριν το επόμενο καλοκαίρι τους αριθμούς αυτούς, έτσι ώστε να υπάρξει μια αίσθηση κανονικότητας Τώρα για την τουρκική πλευρά. Η επανεγκατάσταση συνεχίζεται με το πρόγραμμα 1 προς 1. Αλλά ο συνολικός αριθμός είναι χαμηλός, 2.760. Η εφαρμογή των δυνατοτήτων του Ταμείου για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, 2,2 δις μέχρι τώρα έχουν δοθεί, έχουν αποφασιστεί να δοθούν, 700 εκατομμύρια έχουν δοθεί, μεταξύ των άλλων για σημαντικά προβλήματα όπως το δίκτυο ασφαλείας κοινωνικής πρόνοιας. Ιατρική βοήθεια δηλαδή για τους πρόσφυγες στον τομέα επίσης της εκπαίδευσης και της φροντίδας των παιδιών. Σχετικά με την απελευθέρωση των θεωρήσεων θα είμαι σύντομος, υπάρχουν 7 benchmarks τα οποία ακόμα δεν έχουν καλυφθεί. Σύντομα τώρα για τις ε, συνθήκες που επικρατούν λόγω των εξαιρετικά κακών συνθήκων λόγω κλίματος. Η Ελλάδα χτυπήθηκε τις τελευταίες μέρες από άσχημο καιρό, χειμερινό, και κατέστησε τις συνθήκες τις δύσκολες κατά τις οποίες ζουν οι μετανάστες ακόμα πιο δύσκολες. Η Επιτροπή είναι σε μόνιμη επαφή με όλους τους εμπλεκομένους τοπικές αρχές, δημόσιες αρχές, κοινωνία των πολιτών για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι σημαντικό να γίνει η διάκριση ανάμεσα στην κατάσταση στην ενδοχώρα και στα νησιά. Για να μιλήσω για την κατάσταση στην ενδοχώρα να πω ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι τοπικές αρχές και χρηματοδοτούμενοι από εμά εταίροι έκαναν σημαντικά βήματα προετοιμασίας για τη χειμερινή περίοδο στα πλαίσια του κανονικού χειμώνα αν θέλετε δόθηκε προτεραιότητα στον βορρά και στην δύση όπου οι θερμοκρασίες κατεβαίνουν πάρα πολύ ε, τον χειμώνα. Έχει βελτιωθεί η θέρμανση, η παροχή θερμού ε, και διανοή μέσων γενικά έτσι ώστε να βελτιωθεί η, η συνθήκη κατοικίας ε, διαμονής. Η κατάσταση λοιπόν στην ενδοχώρα, στην υπηρετική χώρα είναι σχετικά ελεγχόμενη. Δεν λέω ότι όλα πάνε τέλεια. Πάντως ε, μπορούμε να πούμε ότι σχετικά η κατάσταση εξελίσσεται με διαχειρίσιμο τρόπο. Αν οι πληροφορίες μας είναι σωστές, υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στους 700 πρόσφυγες μετανάστες που παραμένουν σε κλειστούς χώρους με συνθήκες ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των χειμερινών συνθήκων. Αλλά αυτοί ήδη έχουν ξεκινήσει να μετακινούνται σε θερμότερες και, ε, αποτελε... καλύτερες εγκαταστάσεις. Στα νησιά όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη τώρα. Και αυτό εφαρμόζεται κυρίως, ισχύει κυρίως για τη Λέσβο και για τη Σάμο. Στα άλλα τα νησιά Δεν μπορώ να πω ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αλλά στη Λέρο, Κό και Χίο η κατάσταση ελέγχεται. Όμως στη Μυτιλίνη και στη Σάμο υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι και στα δύο νησιά που καλύπτονται ανεπαρκέστατα και δεν έχουν πολλές φορές καθόλου θέρμανση στις κατοικίες τους και αυτό δεν είναι καθόλου αποδεκτό. Ευτυχώς σήμερα βελτιώνεται η θερμοκρασία, αυξήθηκε λίγο αλλά είναι σαφές ότι υπάρχουν κατεπήγοντα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για τη Λέσβο τώρα έχουν ξεκινήσει κάποιες δράσεις, δράσεις οι οποίες μπορεί να πει κανείς ότι σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και με τη στήριξη τη δική μας και των εταίρων μας έχουν αρχίσει να παίρνουν μέτρα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με διάφορους τρόπους. Πρώτον, αυτοί οι οποίοι εντάσσονται στην κανονική διαδικασία ασύλου μεταφέρονται στην υπηρετική χώρα. Υπάρχει συνεργασία του τοπικού πληθυσμού που δεν ήταν δεδομένο πριν ε, ε, ευρεθούν συμπληρωματικοί αριθμοί ε, δωματίων σε ξενοδοχεία, θα προσθεθούν και άλλα ξενοδοχεία. Uh, Επίσης, πήραμε άδεια επιτέλους για να εγκαταστήσουμε οικίσκους προκατασκευασμένους Uh, is putting additional uh, house uh, prefabricated houses there and as you may have seen in in the press the Όπως είδατε ίσως στο μέσα ενημέρωσης το ελληνικό ναυτικό έστειλε ένα σκάφος μεγάλο και ένα αρματαγωγό και οι πρώτες ομάδες προσφύγων εγκαθίστανται τώρα στο πλοίο ε, γύρω στα 300 άτομα μπορούν να βρουν καταφύγιο εκεί. Στη Λέσβο λοιπόν τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Στη Σάμο είναι οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει συνεργασία για να βρεθούν κατοικίες εκτός των κέντρων των κλειστών και προσπαθούμε να βρούμε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις οι οποίες σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση είναι διαθέσιμες αλλά μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει βρεθεί λύση. Και δεν υπάρχει αρκετός χώρος, οργανωμένος χώρος, όπου να έχουμε την δυνατότητα πλέον να εγκαταστήσουμε τους οικίσκους. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στη Σάμμο λοιπόν, για να βρούμε λύσεις για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι οι χειμερινέ συνθήκες δημιούργησαν περαιτέρω θέματα και έπρεπε να τα αναφέρω. Ο πρόεδρος Μωράης, σας ευχαριστώ για την πρώτη αυτή τοποθέτηση. Ασφαλώς θα υπάρξουν ερωτήσεις. Αν θέλετε να ακούσουμε τον κύριο Ράιαν πρώτα. Μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά γιατί μετά τα πεπειραμένα μέλη μας θα σας υποβάλουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος όσο γι' αυτό γίνεται. Δύο πρόσθετες εκθέσεις που εγκρίθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου πρώτα για μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση, η 8η έκθεση και η τέταρτη σύσταση για την αποκατάσταση των μεταφορών Δουβλίνου στην Ελλάδα. Πρώτα η 8η έκθεση για μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη σχετική έκθεση και για τις δύο αυτές μορφές αλληλεγγύης που εξακολουθούν να αποτελούν ε, κύρια πολιτική προτεραιότητα για να προσφερθεί βοήθεια και στήριξη και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέφερε το θέμα και δήλωσε ότι θα προσφέρει περαιτέρω στήριξη και ιδίω για ασυνόδευτους ανηλίκους. Ο, έγινε κάποια σημαντική πρόοδος στην τελευταία περίοδο του παρελθόντος έτους. Περίπου 1.500 μετεγκαταστάσεις έγιναν τον Νοέμβριο και το υψηλότερο νούμερο μέσα σε περίοδο μηνός. Ο αριθμός των μετεγκαταστάσεων ε, από την Ελλάδα έχουν φτάσει και σταθεροποιηθεί στους χίλιους τον μήνα. Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι μετεγκαταστάσεις και από την Ιταλία πρόσφατα. Τον Νοέμβριο ήταν και το υψηλότερο νούμερο έως τώρα. μέχρι 8.000 άτομα είχαν μετεκατασταθεί μέχρι το Σεπτέμβριο πέρσι. Μέχρι χθε είχαμε ξεπεράσει το κατόφλιο των 10.000, άρα συνεχίζεται αυτή η θετική τάση. Είναι προφανές από τους αριθμούς αυτούς ότι απέχουμε ακόμη πολύ από τα νούμερα για τα οποία είχαν δεσμευτεί οι χώρες μέλη τον Σεπτέμβριο του 2015 είναι σωστό ωστόσο να σημειωθεί ότι η πρόσφατη θετική τάση είναι μια καμπύλη ανερχόμενη και μάλιστα αρκετά απότομα και η δέσμευση για τη μετεκατάσταση ασφαλώς υλοποιείται και αυτό είναι καλό. Τώρα, σαφώς μένουν σημαντικές προσπάθειες να γίνουν για να ξεπεραστούν τα πρακτικά εμπόδια, τα πρακτικά διοικητικά εμπόδια και να αυξηθούν και οι δεσμεύσεις, η προθυμία των χωρών μελών να υποδεχθούν περισσότερα πρόσωπα μέσω του relocation. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σύστασή της έχει προσαρμόσει τους στόχους που θεωρεί ότι είναι ρεαλιστικοί και επιθυμητοί για την μετεγκατάσταση και θεωρούμε ότι είναι δυνατό τώρα να μεταφερθούν όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφοι για μετεκατάσταση από Ελλάδα και Ιταλία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Οπότε και εκπνέει η διαδικασία αυτή και έχουμε βάλει στην σύσταση ρητά ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να στοχεύουν σε μετεγκατάσταση τουλάχιστον 2.000 ατόμων τον μήνα από την Ιταλία και 3.000 από τον Απρίλιο και 2.000 από, το, από την Ιταλία και 1.500 από τον Απρίλιο και μετά. Για να μπορέσουμε να μετεγκαταστήσουμε όλους τους μετεγκαταστήσιμους, ας το πω έτσι, ε, υποβάλλοντες άσυλο, ε, αίτηση ασύλου δηλαδή. Ε, επιτρέψτε μου να μην πω σε όλες τις λεπτομέρειες της εκθέσεως, αλλά πάντως ε, αυτή τονίζει ορισμένα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και κάποιες δράσεις που έχουν γίνει και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες μέλη. Τελευταία, ο κύριος Βέρουεϊ εξήγησε τις προσπάθειες που αναλαμβάνουν οι ελληνικές αρχές για την καταχώρηση. Αυτό διευκολύνει και την διαδικασία μετεγκαταστάσεως και για πρόσωπα δηλαδή που είναι επιλέξιμα. Το ίδιο στην Ιταλία υπάρχει ανάγκη οι Ιταλικές αρχές να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους και να διαθέσουν προσωπικό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 1.500 αναμήνα που είναι ρεαλιστικός. Άλλα βήματα γίνονται για να επιληθούν ορισμένα προβλήματα σχετικά με τον χρόνο που απαιτείται για να γίνουν οι έλεγχοι ασφαλείας στην Ιταλία και με, τον, ε, τη βοήθεια της Ευρωπόλ. Ο αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων που μετεκαθίστανται είναι ακόμη απογοητευτικός, αλλά πάντως έχει γίνει κάποια πρόοδος, 200 περίπου έχουν μετεγκατασταθεί. Από την Ιταλία μόνο ένας μέχρι τώρα. Γίνονται όμως και άλλες προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα νομικά κολλήματα στην Ιταλία, ώστε να μπορέσουν να επαναληφθούν οι μετεγκαταστάσεις όσο γίνεται γρηγορότερα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δεσμεύσεις, τις pledges, Ζητεί βέβαια η έκθεση από τις χώρες μέλη να τις αυξήσουν. Οι standing pledges ήταν 20.000 οι ε, δεσμεύσεις δηλαδή που είχαν αναλυφθεί. Έχει γίνει μια πρόοδο στο μεταξύ. Βέβαια, ζητείται από τις χώρες μέλη να αυξήσουν τις δεσμεύσεις αυτές. Είναι πολύ διαφορετική κατάσταση ένα χώρα μέλος. Ορισμένες χώρες μέλη μόλις και έχουν μετεγκαταστήσει ελαχίστους, ενώ άλλες έχουν ε, ε, υποδεχτεί σημαντικούς αριθμούς. Πολύ σύντομα τώρα για την επανεγκατάσταση εκεί, νομίζω η κατάσταση είναι πιο θετική με την έννοια ότι πάνω από τους μισούς των θέσεων για resettlement που είχαν ε, αποτελέσει το δικείμενο της δέσμευσης τον Ιούλιο, Ιούλιο του 2015 Έχουμε δηλαδή ξεπεράσει 14.000 από τις 22.500 θέσεις που είχαν υποσχεθεί οι χώρες μέλη και ένα σημαντικός αριθμός από Τουρκία, Ιορδανία και Λίβανο και στην περίοδο της εκθέσεως είχαμε ένα αριθμό περίπου 3.000 που επανεκαταστάθηκαν από την Τουρκία. και σύμφωνα και με τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας όπως εξήγησε πριν ο Βερβέη. Αναμένουμε όλες οι δεσμεύσεις για resettlement του Ιουλίου 2015 να υλοποιηθούν μέχρι τέλους του έτους. Αυτά για μετεγκατάσταση και πανεγκατάσταση και τη σχετική έκθεση. Τώρα για την ε, σύσταση Back to Dublin για την Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο γκρίναμε την τέταρτη σύσταση. Οι πρώτες τρεις αναφέρονται μοναχά στην Ελλάδα. Αυτή του Δεκεμβρίου, όχι Σεπτεμβρίου, ε, απευθυνόταν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες μέλη. Πολύ σύντομα υπενθυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε την διαδικασία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι είναι ότι από το 2011 είχαμε στην ουσία αναστολή όλων των μεταφορών Δουβλίνου προς την Ελλάδα και αυτό είχε ένα σημαντικό αρνητικό αποτέλεσμα στη λειτουργία του συστήματος Σέγγεν δημιουργεί και κίνητρα για τους ετούντες άσυλο να μετακινούνται παράνομα και προς άλλες χώρες μέλη και αυτός να κάνουν και δευτερεύουσες μετακινήσεις και επιπροσθέτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταγράψει σημαντικές βελτιώσεις που έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα και ιδίως ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο και το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα Ορισμένες από τις πιο βασικές πτυχές αυτών είναι ότι έχουμε τώρα μια ειδική υπηρεσία ασύλου στην Ελλάδα που τριπλασίασε το στελεχικό δυναμικό της στο τελευταίο χρόνο. Έχουμε και καλύτερες δυνατότητες υποδοχής, σημαντική αύξηση των αριθμών θέσεων σε σύγκριση με έστω και πριν από ένα έτος. Έχουμε σημαντική αύξηση του δυναμικού των επιτροπών προσφυγών, όπως είπε πάλι ο Μάρτιν, και σε ό,τι αφορά το δυναμικό αλλά και την σύνθεση των επιτροπών είδαμε βελτίωση τα, τον τελευταίο χρόνο προς θετική κατεύθυνση επομένως σημαντικά βήματα έγιναν και για το νομικό πλαίσιο στο νομικό πλαίσιο καλύτερα εκκρεμεί Βέβαια, η καθιέρωση ενός πλαισίου που να επιτρέπει δωρεάν νομική αρρωγή προς όλους τους τούντες άσυλο στα ελληνικά νησιά και για τους περισσότερους από αυτούς που βρίσκονται στην υπηρετική Ελλάδα. Όμως, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τονίζει αυτό στην έκθεσή της, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στο σύστημα ασύλου στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα των καταλημάτων. Αυτά εξηγήθηκαν προηγουμένως από τον συνάδελφό μου Βερβέη. Σημαντικό είναι να τονιστεί ακόμη ότι υπάρχουν προβλήματα στην αντιμετώπιση πιο ευάλωτων ε, του άσυλο και ιδίω των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς επίσης προβλήματα σημειώνονται και με την ταχύτητα της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Πριν να έρθω στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τις σημαντικές πιέσεις που υφίσταται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις ε, σημαντικές σε αριθμό αφήξεις, τεράστιο αριθμό αφήξεων στο τέλος του 2015 και αρχές του 2016, τον σημαντικό αριθμό συνεχιζόμενων αφήξεων τις σημαντικές προσπάθειες που εφαρμόζει η Ελλάδα για που καταβάλει μάλλον η Ελλάδα για την εφαρμογή της ε, Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία, το κλείσιμο του βόρειου διαδρόμου από το αρχέ του 2016, την πολύ σημαντική αύξηση της ε, νομολογίας που αντιμετωπίζει η Επιτροπή Ασύλου από τότε που άρχισε το εγχείρημα αυτό το τελευταίο καλοκαίρι και που έχει οδηγήσει στο να αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ασύλου από οποτεδήποτε στο παρελθόν. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Και για τους λόγους αυτούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στη σύσταση να μην προχωρήσουμε σε άμεση πλήρη επανάληψη των μεταφορών Δουβλίνου, αλλά σε σταδιακή επανάληψη. Οι μεταφορές αρχίσουν λοιπόν από την Άνοιξη φέτος αναφορικά με πρόσωπα που φτάνουν στην Ελλάδα από τα μέσα Μαρτίου και μετά επί προσθέτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι ευάλωτοι ετούντες άσυλο δεν θα πρέπει να μεταφέρονται και ένα άλλο σημαντικό είναι ότι δεν θα πρέπει να γίνονται μεταφορές εάν δεν υπάρχουν ειδικέ εξασφαλίσεις από τις ελληνικές αρχές που ακριβώς θα εγγυώνται ότι τα πρόσωπα που θα μεταφερθούν στην Ελλάδα θα τύχουν μεταχείρισης απόλυτα συμμορφούμενης με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ότι θα έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής, ότι οι αιτήσει τους θα αντιμετωπίζονται με ταχύ τρόπο ότι θα καταλήγουν σε ειδικά διαμορφωμένα κέντρα υποδοχής. Προβλέπουμε επίσης ότι ο αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Ασύλου θα παίζει ρόλο στην, στον έλεγχο της συμμόρφωσης και έχουμε αρχίσει ήδη τις συζητήσεις με την ΕΑΣΟ για το πώς θα συμβεί αυτό. Θα είμαστε βέβαια σε πολύ στενή διασύνδεση με τις ελληνικές αρχές για όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να μας αναφέρουν περί τα μέσα Φεβρουαρίου για τα περαιτέρω βήματα που εμείς έχουμε συστήσει ότι θα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των εκκρεμουσών ελήψεων στο σύστημα ασύλου, να μας εξηγήσουν και πώς ακριβώς θα ε, δοθούν οι εγγύησεις που ζητούμε και θα υποβάλουν μετά αναφορές αναδίμηνο Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αυτό είναι σαφές. Ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες πιέσεις θα αντιμετωπίσει ακόμη η Ελλάδα τους επόμενους μήνες ή χρόνια. Γι' αυτό στην σύστασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι θα παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και αν χρειαστεί να υποβάλουμε νέες συστάσεις ή διευκρινήσεις επί των συστάσεων που έχουμε ήδη κάνει, ως, όπως αυτό μπορεί να θεωρηθεί, όπως θα θεωρηθεί αναλόγως αναγκαίο. Ε, και ένα τελευταίο αλλά σημαντικό που πρέπει νομίζω να τονιστεί είναι ότι η σύσταση τονίζει ένα θέμα κάπως πολιτικού χαρακτήρα ότι οι υποχρώσεις δεν βαρύνουν μόνο την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες μέλη σε ό,τι αφορά την στήριξη που προσφέρουν στην Ελλάδα και σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των δεσμεύσεών τους για με την κατάσταση που έχουν κάνει ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 και τα είπα αυτά πριν, αλλά και κάτι σημαντικό που νομίζω ανέφερε και ο Μάρτιν όσον αφορά την αποστολή εμπειρογνωμόνων στην ΕΑΣΟ που θα βοηθήσουν με τη σειρά τους τις ελληνικές αρχές τις σημαντικές προσπάθειες που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση εκεί και ιδίως στα ελληνικά νησιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Χαίρομαι που εξετάσαμε αυτό το ζήτημα σήμερα. Παρότι δεν έχουμε αθρώα προσέλευση, αλλά ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήρθαν. Η κυρία Γετυπέρη έχει πρώτο λόγο. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Έχω ορισμένα θέματα. Κάποιε φορέ αφορούν μόνο την ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, άλλε ε, αφορούν τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ότι το Σεπτέμβριο του 2015 υπήρχε ήδη κάποια προετοιμασία για τον χειμώνα, συμφωνία αύξηση ε, τη χωρητικότητα υποδοχή και ε, με κινητοποίηση του μηχανισμού πολιτική Προστασία, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ρωτώ λοιπόν αν έχει γίνει αυτό, ότι η Ελλάδα θα ε, αυξήσει την ε, δυνατότητα υποδοχή στι 20.000 θέσει. Τι συνέβη λοιπόν με αυτές τις μεγάλες ε, δηλώσεις και διακηρύξεις του Σεπτέμβριο του 2015 και μετά αν δούμε τη Βαλκανική Οδό και πάλι έχουμε απαράδεκτες εικόνες από τη Σερβία η πρώτη του ΟΗΕ για του Πρόσφυγε θα αύξανε στι 50.000 θέσει στη χωρητικότητα αποδοχής. Δεν κατανοώ λοιπόν γιατί οι άνθρωποι κοιμούνται έξω στο δρόμο σε τόσο ε, άσχημες καιρικές συνθήκες. Τι συνέβη λοιπόν με όλες αυτές τις διακηρύξεις που είχαν παρουσιαστεί ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 ως μια συμφωνία. Κάτι το οποίο είχε ήδη δηλαδή λυθεί. Μετά για τον κύριο Βερβέ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο γιατί όταν υπάρχει συμφωνία με, τη συμφωνία με την Τουρκία επανεισδοχής να μπορούμε να στείλουμε πίσω και αυτούς που δεν χρήζουν του καθεστώτος του πρόσφυγα. Αυτό ισχύει και για, τους, για όσους υπάρχουν στα νησιά. Γιατί μετά από δύο μήνες είδαμε ότι οι επιστροφές έχουν σταματήσει σχεδόν ολοκληρωτικά. 800 άτομα είδα το προηγούμενο διάστημα, 400 το πρώτο δίμηνο και μετά σχεδόν σταμάτησαν. Αυτές, τι συνέβη όμως τώρα, αυτές οι, με τις, τις χειμερινές συνθήκες, έχετε κάνει κάτι παραπάνω. Προς τον κύριο Ράιαν για την μετακατάσταση. Είναι σχεδόν ένα μαθηματικό πρότυπο. Ε, τόσες δεσμεύσεις έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Αν ε, το διαιρέσουμε με τον αριθμό των μηνών, έχουμε 3.500 από τον Μάρτιο και μετά για τη μετακατάσταση από την Ελλάδα και 1.000, αν κατάλαβα καλά, από την Ιταλία. Όμως, τι θα αλλάξει τώρα. Κατανοώ θεωρητικά και με το μαθηματικό τύπο πώς θα καταλήξουμε στο συνολικό ρυθμό μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά δεν κατανοώ τι θα αλλάξει και τι αυτό που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή ξαφνικά θα αρχίσει να συμβαίνει. Και σε μεγάλη κλίμακα κιόλα. Τέλο. Για την επανεγκατάσταση στην Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, η πρώτη πρόταση και η πρώτη δέσμευση την οποία αναλαμβάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτε είναι να αντικαταστήσουν την παράνομη οδό με μία νόμιμη. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου βλέπουμε ότι αυτό το κομμάτι έχει διαγραφεί. Όμω αυτό είναι το πρώτο σημείο στην Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Επομένω, γιατί είναι επανεγκατάσταση ένα ερώτημα. Συμφωνήθηκε πέραν από το ένα προ έναν. Έχουμε τον αριθμό των παράνομων που φτάνουν στα νησιά ότι θα φτιάχναμε και ένα μεγάλο ε, πρόγραμμα επανεγκατάστασης τι συμβαίνει όμως εκεί, γιατί ακόμα δεν υπάρχει νόμιμη οδός. Και τέλος, και πάλι προς τον κύριο Ράιεν, είπατε ε, μία απίστευτη δήλωση του Επιτρόπου Απραμόπουλου ότι από την 1η Μαρτίου θα πρέπει να ξεκινήσουν και πάλι οι επιστροφές ε, υπό το Δουβλίνο. Τώρα, ρεαλιστικά αν δούμε τα πράγματα, βλέπουμε τις εικόνες από την Ελλάδα και εσείς ο ίδιος αναφέρατε όλα τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμα. Δεν, δεν στέλνουμε εδώ και χρόνια κόσμο πίσω στην Ελλάδα. Όχι από πέρσι. Γιατί ακριβώ δεν υπήρχαν κατάλληλα συνθήκε υποδοχή. Νομίζω και φοβάμαι ότι τροφοδοτείται το λαϊκισμό όταν ανακοινώνεται κάτι που όλοι εδώ ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Ευχαριστώ πολύ, Κίτη. Θα ακούσουμε όλες ε, τις παρατηρήσεις πριν ε, δώσουμε και πάλι το λόγο ε, στους δύο Η κυρία Γκόμες, παρακαλώ. Ευχαριστώ που μας είπατε ότι ο αριθμός ε, των επιστροφών υπό αυτή την ε, ανήθικη και παράνομη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας είναι μόλις 1.240 ε, άνθρωποι από τον Μάρτιο του 2016. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί από μας σας είπαν, σε εσάς δηλαδή την Επιτροπή, και είπαν και σε όσους κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία ότι είναι και μη αποτελεσματική, όχι μόνο παράνομη και ανήθικη, είναι και αναποτελεσματική. Θα ήθελα να επισημάνω αυτό που είπατε και γνωρίζουμε και εμείς από τις ε, εικόνες που έχουμε δει. Τα hot spots στην Ελλάδα. Εξαιτία των άθλων συνθήκων ε, διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν προβληματίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, επιπτώσεις ως προς τη ριζοσπαστικοποίηση ότι θα δημιουργήσει δυσανασχέτιση και μίσος. Εγώ αν ήμουν μεταξύ αυτών των ετούντων άσυλο, θα ήμουν εξαιρετικά εξοργισμένη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που μου συμπεριφέρεται με τόσο παράδεκτο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον, δεν ανησυχεί πώς αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί ε, και για την προπαγάνδα και για τη ριζοσπαστικοποίηση. Τι κάνει λοιπόν η Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ε, επανεγκατάσταση. Εδώ έχουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτών των ε, ε, Γεζίντι που μας απασχολεί από τον Απρίλιο πέρσι και εμένα και τους συναδέλφους. Πέρσι τον Νοέμβριο πήγαμε στην Ελλάδα και είδαμε ότι 600 από τους 1.800 ανθρώπους είχαν καταγραφεί αλλά ούτε ένα όνομα δεν είχε υποβληθεί στα, στις χώρες ε, που ήταν διατεθειμένες να τους υποδεχθούν όπως η Πορτογαλία. Μετά έφτασαν 100 ονόματα. Ακόμα εκεί βρίσκονται όμως αυτά τα άτομα υπό άθλες συνθήκες. Τι κάνει λοιπόν η Κομισιόν για να ε, διευθετήσει αυτό το ζήτημα. Αποδεχόμαστε ότι αυτή η γεζίτη είναι θύματα γενοκτονίας. Γιατί λοιπόν επιτρέπουμε τη συνέχιση αυτής της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης αντί να επιταχύνουμε τη διαδικασία επανεκατάστασής τους. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τούτου. Έχουμε γράψει σε όλους. Στην Επιτροπή, σε όλους τους επιτρόπους. Τίποτα δεν έχει συμβεί. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και τέλος, είχαμε σήμερα εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί και για άλλα κύματα. Δεν αποκλείεται. Να έχουμε πολύ μεγαλύτερες ροές στο μέλλον. Τι είδους προετοιμασίες κάνετε αυτή τη στιγμή, τι κάνετε για αυτούς που αποκαλούμε ασυνόδευτους ανηλίκους, αλλά είναι παιδιά. Έτσι πρέπει να φερόμαστε και όχι να τους αφήνουμε στην τύχη τους και να εξαφανίζονται ε, και τελικά να καταλήγουν σε διάφορα εγκληματικά δίκτυα προς εκμετάλλευση και κακοποίησή τους. Βλέπουμε αυτές τις τρομερές εικόνες από τη Σερβία και από αλλού, όπως είπε συνάδελφος, Πολύ φοβάμαι ότι οι κυβερνήσει μας και τα θεσμικά μας όργανα ε, τροφοδοτούν ε, τον λαϊκισμό και τα ακόμα χειρότερα ε, που συνεπάγει το λαϊκισμός. Ευχαριστώ κυρία Σαρτιντίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κατάσταση στους καταβλισμούς στην Ελλάδα δεν είναι ιδανική. Εντάξει, έχουμε τον εφημισμό, αλλά υπάρχουν και όρια στους εφημισμούς. Δεν γίνεται να λέτε ότι είναι κάτι λιγότερο από ιδανικός είμαι στις 5.30 εδώ και όχι στο τρένο για το Άμστανταμ. Αυτό δεν είναι ιδανικό. Αλλά το να βρίσκεται κανείς σε μία ε, σκηνή, σε ένα καταβλισμό κάπου και ε, να ε, βιώνει αυτές τις άθλιες καιρικέ συνθήκες, όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι λιγότερο από ιδανικό. Είναι ο εφημισμός από τη μία και από την άλλη έχουμε και τους ευσεβείς πόθους ό,τι αφορά τις, τους ρυθμούς επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης. Αυτό είναι κάτι άλλο. Λέτε συνεχώ ότι εξαιτία τη ε, συμφωνία με την Τουρκία ο αριθμό ε, των μεταναστών που έφτασαν στα νησιά έχει πέσει δραματικά. Δεν ισχύει τα στοιχεία και από την υπατηρμοστή του ΟΗΕ δείχνουν ότι το Νοέμβριο του 2015 υπήρχε ε, μια σταδιακή και σταθερή μείωση. Με μια μικρή αύξηση και πάλι δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της συμφωνία, αλλά από τον Νοέμβριο είχαμε πτωτική τάση, όταν οι χώρες στη Βαλκανική Οδό άρχισαν να κλείνουν τα σύνορα. Αυτή η τάση υπήρχε από τον Νοέμβριο του 2015 και υπενθυμίζω ο ε, Υπουργό ε, ε, Μετανάστευση τη Ολλανδία είπε ότι είτε ισχύσει ε, η συμφωνία με την Τουρκία είτε όχι, έχει κλείσει η Βαλκανική Οδό και αυτό θα μα βοηθήσει πολύ. Δεν μου αρέσει που χρησιμοποιούμε το παράδειγμα της συμφωνίας με την Τουρκία ως παράδειγμα για άλλες περιπτώσεις. Ο Πρωθυπουργό τη Μάλτα ξεκίνησε με την Προεδρία και ανέφερε ε, τι καλή που είναι η συμφωνία με την Τουρκία και πώ μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλε ε, περιοχέ. Αυτό είναι πρόβλημα. Τώρα, θα ήθελα διευκρινήσει σε κάτι που ανέφερε αξιωματούχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μία συνεδρίαση τη ε, Σοφίντ Φελτ για την ε, οδηγία υποδοχή. Εκεί αναφέρθηκε λοιπόν ότι οι Τούρκοι ερμήνευσαν την συμφωνία με την Τουρκία ω εξή. Ότι παίρνουν πίσω κάποιον στον κανένα ένα προς έναν όταν είναι ακόμα στα νησιά. Και η Επιτροπή είπε ότι αυτό είναι ο λόγο που οι άνθρωποι δεν προχωρούν από τα νησιά να περάσουν στην ενδοχώρα. Ισχύει αυτό. Μπορούμε να το λάβουμε γραπτό. Θα ήθελα να καταλάβω επιτέλου τη συμφωνία με την Τουρκία. Γιατί κρατάμε του ανθρώπου υπό άθλιε συνθήκε στα νησιά, γιατί δάλου δεν θα του πάρει πίσω η Τουρκία. Γιατί τότε τα πράγματα είναι λίγο ύποπτα, έτσι δεν είναι. Τώρα για τις επιστροφές από το Δουβλίνο από, από το Μάρτιο και μετά. Μόνο αυτοί που έχουν φτάσει από το Μάρτιο, φτάνουν μάλλον το Μάρτιο του 2017 και μετά. Μιλάμε λοιπόν κάποια στιγμή το καλοκαίρι, αργότερα, μέσα στη χρονιά, κάποια άτομα που ενδέχεται να θεωρηθεί ότι μπορούν να επιστραφούν προς την Ελλάδα. Γιατί το κάνουμε και του δίνουμε τέτοιες διαστάσεις ε, δημοσίευσης. Αυτό το αφήγημα δεν βοηθάει κανέναν, ούτε την Ελλάδα, ούτε τους ε, Ευρωπαίους πολίτες και νομίζω ότι κάτι πήρε έχει δίκιο όταν λέει ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Γιατί μετά και πάλι θα υπάρξει υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου που θα λέει η κατάσταση στην Ελλάδα δεν έχει αλλάξει σχέση με πριν από μερικά χρόνια, δεν ε, συμμορφούνται με ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, είναι απάνθρωπο να επιστρέφονται άνθρωποι στην Ελλάδα και ξεκινάμε από την αρχή. Το ξέρουμε, το βλέπουμε, βλέπουμε ότι εκεί θα πάνε τα πράγματα, γιατί κάνουμε λοιπόν αυτή την πρόταση. Εμείς στην Ολλανδία στέλνουμε πίσω ε, ετούντες προς τη Γερμανία. Δεν είμαστε σωστοί ο ένας απέναντι στον άλλον και δεν βοηθάει κανέναν. ...2.007 άτομα είπατε ότι έχουν επανεγκατασταθεί προς την Τουρκία. Πού είναι οι νόμιμες οδοί όμως... Και έτσι κι αλλιώς είχαμε αναφέρει ότι 20.000 άτομα θα ε, περνούσαν από την επανεγκατάσταση. Αλλά τα 2007 άμα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγαμε ότι τα άτομα αυτά βλέπουν νόημα να παραμείνουν στους καταβλισμούς στην Τουρκία. Γιατί δεν είναι θέμα οικονομικό, ε, είναι ε, θέμα ε, του μέλλοντος των παιδιών μας. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πώς γίνεται να είναι τόσο χαμηλά τα αριθμητικά στοιχεία δεν ε, γίνεται να αιτιολογείται μόνο από αυτό που προανέφερα ότι πρέπει να είναι στα νησιά ε, αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, οι εφημισμοί και οι ευσεβείς πόθη δεν θα μας δώσουν καμία λύση σε αυτή την ε, προσφυγική και μάλλον πολιτική, θα έλεγα, κρίση. Ευχαριστώ, κύριε Λενάρτς. Thank you, thank you very much. Σας ευχαριστώ, φίλε Πρόεδρε. Ποτέ δεν θα έλεγα ότι η παρουσία της κυρίας Αργεντίνη θα ήταν sub-optimal στην ε, αίθουσα εδώ. Μπορεί να συζητήσει κανείς αν η συμφωνία με την Τουρκία ή το κρίσιμο της Βαλκανικής Οδού ήταν ο πραγματικός λόγος για τη μείωση των αφήξεων. Κάτι όμως που είναι πέραν συζητήσεως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που πνίγηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, τη μείωσή του δηλαδή του αριθμού αυτού, της ίδιας συμφωνίας. Και ίσως αυτό να είναι ένα παράδειγμα που θα προκύψει και από άλλες συμφωνίες του μέλλοντος, ειδικά για τη Μεσόγειο. Εδώ πράγματι διαφωνούμε για την αξία της τουρκικής συμφωνίας. Υπάρχει πάντως συμφωνία με την Τουρκία, υπάρχει το σύστημα αυτό, τουλάχιστον να φροντίσουμε οι συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί το σύστημα και εκτελεί τη συμφωνία να είναι optimal. Και διαβάζοντας και σε άλλες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχουμε στα νησιά 16.000 άτομα ενώ είναι μόνο 8.000 θέσεις ότι υπάρχουν και μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν ε, απαρκές κατάλημα, ότι δεν υπάρχουν ε, εγκαταστάσεις υγιεινής μέσα στο χειμώνα και, όλα αυτά. Αν θέλουμε να λειτουργήσει η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας θα πρέπει τουλάχιστον να φροντίσουμε οι συνθήκες υποδοχής και εγκατάστασης των ε, ε, προσφύγων και μεταναστών να είναι ασφαλώς πάρα πολύ καλύτερες. Και πριν αρχίσουμε τις επαναφορές στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν βελτιωθεί πολύ σημαντικά οι συνθήκες γιατί τελείως δεν είναι καν ρεαλιστικό να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε να στέλνουμε ανθρώπους ξανά στην Ελλάδα υπό την ισχύ των διατάξεων του Δουβλίνου. Δεν ξέρω αν είναι νομικά δυνατό αυτό που θα ρωτήσω τώρα, αλλά μήπως είναι δυνατό να καταστήσουμε δυνατό αυτό για τις χώρες εκείνες μέλη μόνον οι οποίες έχουν ήδη υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τους για τις επανεγκαταστάσεις ή μετεγκαταστάσεις διότι τον Σεπτέμβριο του 2017 θα έχουμε τα δύο χρόνια και αν κάνω ένα σύντομο υπολογισμό σύμφωνα και με τις συστάσεις και με το ρυθμό των μετεγκαταστάσεων που αναφέρατε προηγουμένως θα έχουμε φτάσει περίπου στις 33.000 περίπου άτομα το Σεπτέμβριο του 2017 ξαναλέω ενώ προβλεπόταν αρχικά γύρω στις 100.000. Και νομίζω είπατε ακόμη ότι εάν συνεχίσουμε με το ρυθμό αυτό, άνθρωποι που είναι επιλέξιμοι για μετεγκατάσταση θα μετεκαθίστανται και η διαφορά μεταξύ, ανάμεσα μάλλον 33.000 και 100.000, πού βρίσκεται. Ή μήπως έγινε λάθος υπολογισμός των επιλέξιμων για μετεγκατάσταση ή υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ιταλία και στην Ελλάδα που δεν τους θεωρούμε επιλέξιμους για μετεγκατάσταση. Ευχαριστώ. Λάμπερτς. Η Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ ερωτήσεις. Πρώτα, συντονισμός. Ακούμε ότι το ΕΚΟ είναι λειτουργικό, ο ύπατο αμοστή για του πρόσφυγε είναι, υπο, λειτουργικός, η ελληνική κυβέρνηση είναι λειτουργική. Ποια είναι η συνεργασία, Ποιο είναι ο συντονισμός ανάμεσα στις αρχές αυτές. Γνωρίζουμε ότι είναι συμπληρωματικό ο χαρακτήρας του έργου τους και όχι επικαλυπτικός. Καλύπτονται τα κενά όμω, διότι από ορισμένα από τα πράγματα που ακούμε φαίνεται ότι ό,τι υπόμνημα συνεννόησης και να υπάρχει δεν αποδίδει υπέρ είτε της ίδιας της Ελλάδος και, πάντοτε, και πάντως σίγουρα όχι υπέρ των ετούντων άσυλο. Ένα από τα πράγματα που έχουμε ζητήσει εξ αρχής από το Κοινοβούλιο, εμείς εδώ του Κοινοβουλίου δηλαδή, είναι η μετακίνηση των ανθρώπων από τα νησιά, όπου ασφαλώς υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυσκολίες, όπως άλλωστε εξηγήθηκαν και προηγουμένως, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές δυσκολίες ξεχάστε την, ε, ε, τις ε, πραγματικές περιστάσεις ε, της υποδοχής. Για να μετακινηθούν στην υπηρετική χώρα θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικό να εγκαθίσταται οι άνθρωποι αυτοί σε τόπους χωρίς θέρμανση σε πρώην εργοστάσιο πυρομαχικών που δεν έχει απολύτως τίποτα μέσα. χημικά εργοστάσια, πάλι χωρίς θέρμανση, με κατάλοιπα ενδεχομένω από τις ουσίες που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή πυρομαχικών και χημικών ουσιών κτλ. Κάπου υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που λειτουργούν, αλλού όχι. Γνωρίζουμε ποια είναι και τα προβλήματα των ε, ελληνικών υπηρεσιών υγείας Γνωρίζουμε ποιε είναι οι πιέσει που αντιμετωπίζει το ελληνικό σύστημα υγεία και δεν μιλώ καν γι' αυτό. Είστε ικανοποιημένοι, εσεί είμαστε ικανοποιημένε, εμεί, ότι οι πόροι που χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται επαρκώ ώστε να προσφέρουν μια βασική κάλυψη στου ανθρώπου αυτού. Και ό,τι δεν υπάρχει, προσπαθούμε να καλύψουμε. Καλύπτουμε τα κενά. Υπάρχουν χώρε μέλη οι οποίε παρεμβαίνουν για να στηρίξουν ώστε να επιταχυνθεί η μετεγκατάσταση. Γνωρίζουμε όσα γνωρίζουμε για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ή με σταυρωμένα χέρια οι χώρες μέλη, διότι στηρίζονται στην βάση ότι Ε, εν πάση περιπτώσει πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να ε, υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας ή απλώς αφήνουμε τον κόσμο εκεί να σαπίζει. Τα χρήματα που δαπανώνται στην Ελλάδα και τα ποσά φαίνονται σημαντικά. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι ικανοποιητική η, η χνηλάτιση του χρήματος αυτού. Πού πηγαίνουν δηλαδή τα χρήματα αυτά. Ή μήπως υπάρχουν φόβοι ότι κάποια χρήματα χάνονται. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την διαδικασία υποδοχής των φθάνων στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επεστράφησαν που έχουν οικογένειες ή που ισχυρίζονται ότι έχουν οικογένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την ισχύ των διατάξεων του Δουβλίνου θα έπρεπε κανονικά να έχουν το δικαίωμα να ενωθούν με τις οικογένειές τους. Και όμως επεστράφησαν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ε, διαδικασία, την admissibility procedure, μπορούμε να έχουμε διαβεβαίωση ότι όταν θα αρχίσει η διαδικασία του ασύλου, όταν θα λαμβάνονται αποφάσεις για την, ε, ε, για είσοδό τους, θα μπλοκάρονται οι άνθρωποι αυτοί από το να ε, ζητήσουν να ισχύσουν τα δικαιώματά τους που έχουν από το δίκαιο του ασύλου. Για Βάινμπεργκ, εκτός αν υπάρχει κανείς άλλος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τώρα για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας δεν λειτουργήσε εξ αρχής όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι. Εμείς είπαμε ότι η πλειοψηφία των βουλευτών ήταν κατά τη συμφωνίας αυτής βασικά γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Χάνονται δισεκατομμύρια προς όφελος υποσχέσεων. Τι γίνεται λοιπόν με τον εκβιασμό τον οποίο ασκεί η Τουρκία εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μείωση μεταναστών, αλλά υπάρχουν και άλλα, θα έλεγα, δίκτυα, άλλες ροές οι οποίες ενεργοποιούνται. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση, σαν παράδειγμα, των ανθρώπων που θέλουν από την Αφρική να έρθουν στην Ευρώπη μέσω εναλλακτικών οδών. Λοιπόν, η συμφωνία που θα κάνουμε με τη Λιβύη θα είναι το επόμενο στάδιο και με ποιες άλλες χώρες θα υπογράψουμε τέτοιου είδους απαράδεκτες συμφωνίες. Νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, πρέπει να προλάβουμε αυτά τα οποία προμηνύονται διότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται απροετοίμαστη. Πάντως η συμφωνία αυτή δεν είναι συμφωνία, είναι εκβιασμός εις βάρος της Ένωσης από την Τουρκία. Τώρα το θέμα της μετεγκατάστασης αναφέρθηκε από άλλους συναδέλφους. Οι, αριθμοί τους οποίους μας παρουσιάσατε από τον Απρίλιο 3.000 έχουν ε, φύγει από την Ελλάδα και άλλες 3 από την Ιταλία. Νομίζω ότι οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν μια κάποια αύξηση και αυτό δεν είναι κακό. Αλλά έχετε συζητήσει λίγο τις απαιτούμενες διευκρινήσεις για την υποδοχή των μεταναστών αυτών. Για το Δουβλίνο και την Ελλάδα και την επιστροφή στην Ελλάδα. Εδώ και έξι χρόνια οι συζητήσεις αυτές είχαν ήδη γίνει για την ε, ειδική άδεια να μην ε, στέλνονται πίσω οι άνθρωποι αυτοί. Η Ελλάδα υποτίθεται ότι είχε χρόνο για να βελτιώσει την κατάσταση. Τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στους δύο προσκεκλημένους μας. Okay. Uh, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Να ξεκινήσω με το τι έγινε με τις υποσχέσεις οι οποίες είχαν δοθεί το 2015 για την υποδοχή μεταναστών και προσφύγων. Η Ελλάδα τότε είχε αναλάβει την υποχρέωση για τη δημιουργία 30.000 θέσεων και 20.000 η ύπατη αρμοστία. Να πω ότι μέχρι τώρα η Ελλάδα έχει δημιουργήσει πάνω από 15, 55.000, ε, συγγνώμη, 55.000 θέσεις και επίσης και 20.000 από πλευράς της ύπατης αρμοστίας είναι πλέον διαθέσιμες. Συνεπώς λοιπόν η Ελλάδα έχει κάνει πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο αναμένεται τότε. Τότε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας ενεργοποιήθηκε το 2015 και γι' αυτό ε, διετέθησαν σκηνές, οικίσκη κτλ. Η χρηματοδότηση για αυτές τις δραστηριότητες αυξήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια να πω ότι η ΕΚΟ μέχρι τώρα μέσω των εταίρων της έχουν λάβει πάνω από 200, 200 ε, εκατομμύρια. Έχουμε δώσει 350 κατεπίγουσα βοήθεια, ε, είτε άμεσα στο κράτος, είτε σε ε, ανθρωπιστικές οργανώσεις. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι στην παρούσα φάση η έλλειψη υλικού εξοπλισμού προσωπικού κτλ. δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Όπως είπα ότι στην υπηρετική χώρα, όχι ότι όλα είναι καλά πια, αλλά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Το πρόβλημα όμως στα νησιά παραμένει. Έχουμε έλλειψη χώρων στα νησιά διεκδικούμε ήδη από το Μάρτιο του 2016 μεγαλύτερο χώρο υποδοχής. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δυστυχώς υπάρχει πολύ σημαντική τοπική αντίδραση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Υπάρχουν βέβαια δωμάτια ξενοδοχείων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούνται, αλλά απαιτείται προετοιμασία. Δεν θέλω να μιλάω για θέματα που δεν ξέρω πολύ καλά. Για την Βαλκανική οδό, ας πούμε, δεν μπορώ να απαντήσω, διότι δεν είμαι ενημέρος. Τώρα, ε, γιατί οι μη πρόσφυγες δεν επιστρέφονται. Κοιτάξτε, ε, αυτό εξαρτάται από το νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει στην Ευρώπη πριν καθορίσει κανείς αν κάποιος είναι πρόσφυγας ή περνάει από μία συνέντευξη, μπορεί μετά να ασκήσει έφεση και αυτό απαιτεί χρόνο. Το θέμα λοιπόν είναι περισσότερο θέμα χρονισμού παρά οτιδήποτε άλλο. Για νομικούς λοιπόν λόγους κυρίως είναι δύσκολο να επιστρέφουν γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί, να επαναπροωθούνται ταχύτατα. Η αστυνομία έχει κάποια δυσκολία για την έβρεση των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι αναζητούνται για να υπάρξει λοιπόν μια αποτελεσματική πολιτική επαναπροώθησης απαιτούνται οργανωτικές ικανότητες οι οποίες ελείπουν. Υπάρχουν τοπικές αντιδράσεις. Είναι απαραίτητο όμως και για την προστασία των πραγματικών μεταναστών, των, προς, των πραγματικών, των αληθινών προσφύγων, να προχωρήσουμε στην εκαθάρισε. Τώρα η ΕΚΟ, εγώ δεν εκπροσωπώ την ΕΚΟ, αλλά γνωρίζω γιατί συνεργάζομαι μαζί τους. ότι χρηματοδοτούν τοπικούς εταίρους, έχουν συντονιστεί με το Υπουργείο Μετανάστευσης, τέθηκαν πολλά ερωτηματικά για το ποιος κάνει τι, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά. Το θέμα δεν είναι να κρυφτεί κανείς από τις ευθύνες του. Το θέμα δεν είναι η έλλειψη εξοπλισμού, δεν είναι η έλλειψη υλικού, δεν είναι η έλλειψη χρημάτων. Απαιτείται χώρος για να βάλουμε το κυβότο ε, εμπορευματοκιβώτιο ή κάποιες άλλες εγκαταστάσεις. Προσπαθούμε να βρούμε χώρο για να το κάνουμε. Υπήρξαν και αρκετές ε, δηλώσεις, σχόλια, ισχυρισμοί, τα οποία δεν καλούμε να σχολιάσω. Δεν έχω την ψευδέστηση ότι θα σας πείσω για κάτι το διαφορετικό σας αυτά, αυτά τα οποία είπατε. Να πω όμως για το να πούμε τι είναι νόμιμο και τι είναι μη νόμιμο, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς. Εγώ σας παρουσίασα την κατάσταση. Δεν την εφήβρα εγώ την κατάσταση. Καθένας που ζητά άσυλο έχει την δυνατότητα να κάνει αίτηση, να περάσει από συνέντευξη, να έχει συνδρομή, να μπορεί να καταθέσει έφεση, πολλοί το κάνουν αυτό και πολλοί από αυτούς, να είμαι ειλικρινής, παραμένουν στα νησιά. Το να πούμε ότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο, κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι είναι ένας χαρακτηρισμός τον οποίο εγώ μπορώ να κάνω. Παραμένουμε στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Τώρα, για την μετεγκατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση. Δεν θέλω εγώ να δακτυλοδείξω κάποια από τις χώρες, αλλά ο βασικός λόγος για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, γιατί δηλαδή απαιτείται χρόνος για την μετακίνηση και την μετεγκατάσταση και μετά από την αποδοχή τους από τα κράτη-μέλη, είναι γιατί ορισμένες χώρες, και δεν λέω ποιες είναι, μας λένε συνεχεία περιμένετε μια στιγμή, μη μας το στείλετε ακόμα, γιατί πρέπει να προετοιμάσουμε τα της υποδοχής. Υπάρχει λοιπόν μια κάποια συμφωνία επίσημη έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγκατάσταση σε δίμηνο, αυτό δεν ισχύει. Αλλά αυτό δεν οφείλεται στην ελληνική υπηρεσία ασύλου, αυτό οφείλεται στις χώρες μέλη που δεν τους υποδέχονται. Then, um, now, yet another proof that, that Εγώ βέβαια δεν έχω πολιτικές φιλοδοξίες, γιατί από ό,τι φαίνεται πρέπει κάποιος ε, να μιλάει έτσι με τέτοιου είδους ε, σχήματα, όπως η υπερβολή. Εγώ ασχολούμαι με αλλά προσπαθώ να μην υπερβάλλω. Και ζητώ συγγνώμη αν προσβάλλω κάποιον. Το ανέφερα και εγώ προηγουμένως ότι όταν είπα suboptimal, δηλαδή λιγότερο από ιδανικό, το ανέφερα και εγώ έτσι λίγο ηρωνικά. Δεν είμαι πολιτικός βέβαια. Τώρα, κατά πόσο ήταν η συμφωνία με την Τουρκία ή κάτι άλλο που μείωσε τον αριθμό των αφήξεων. Μπορώ να σας στείλω ένα γράφημα που είναι ξεκάθαρο. Σε αντίθεση με τα όσα λέτε, οι αφήξει στους μήνες Νοέμβρη-Δεκέμβρη έως και αρχές Μαρτίου ήταν εξαιρετικά υψηλές. Εξαιρετικά υψηλό ο ρυθμός των αφήξεων. Όντω, έπεσαν οι αφήξει γιατί ήμασταν ε, κατά του χειμερινού μήνε. Όμω, για αυτή την περίοδο, κατά μέσο όρο, για του μήνε που αναφέρατε, έχουμε περίπου 4.000 άτομα κάθε μέρα που κατέφθαναν στα νησιά. Στις εβδομάδες πριν από την κοινή δήλωση με την Τουρκία και πάλι είχαμε 1.700 αφήξεις ανά ημέρα. Την πρώτη μέρα μετά τη δήλωση και πάλι είχαμε 1.600, δεύτερη μέρα 500 και νομίζω ότι μετά πέσαμε στους 250. Και πολύ γρήγορα πέσαμε κάτω από τους 50 την ημέρα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσο είναι ηθική ή όχι συμφωνία, όμως για μένα αδιαφυσβήτητα η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είχε τεράστια επίπτωση στον αριθμό των ε, αφήξεων. Και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ε, σε ό,τι αφορά την αξία της ε, συμφωνίας. Μετά ρωτήσατε κατά πόσο μπορούν αυτά τα άτομα να μεταφερθούν ε, στην υπηρετική Ελλάδα. Ε, συμβαίνει ήδη αυτό και σημαντικό είναι να το αναφέρουμε ότι ήδη μεταφέρονται αυτά τα άτομα ε, στην υπηρετική Ελλάδα. Όμως πρόκειται για άτομα όπου οι αρμόδιες αρχές έχουν θεωρήσει ότι είτε πρόκειται για ευάλωτα άτομα, είτε για λόγους οικογενειακής επανένωσης, δεν θα επιστραφούν στην Τουρκία. Και νομίζω ότι απαντώ έτσι και σε άλλο ερώτημα που αναφέρθηκε προηγουμένως. Τους τελευταίους μήνες περίπου 3.500 άτομα έχουν μεταφερθεί στην υπηρετική Ελλάδα. και υπό τις ισχύουσες συνθήκες κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου όσοι μπορούν να μεταφερθούν και δεν έχουν λόγο να μένουν στα νησιά να μεταφέρονται. Τώρα, για παράδειγμα, όχι οι πρόσφυγες αλλά οι μετανάστες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης η Τουρκία όντως είπε ότι εμείς θα πάρουμε πίσω μόνο άτομα ε, που είναι αυτή τη στιγμή στα νησιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κυρία Σατζεντίνη. Βεβαίως, τα έγγραφα θα λένε ότι κάποιος καταφτάνει σε ένα νησί. Γιατί να μην φτάνει αυτό. Γιατί μιλούμε για περιορισμό στο χώρο, στα νησιά, συμφωνώ απολύτως, αλλά ε, δεν πάμε να πούμε ότι είναι πιο εύκολο να τους κρατήσουμε στα νησιά αντί να τους περάσουμε στην υπηρετική χώρα. Αν πει η Τουρκία θα δεχθώ μόνο τα άτομα ε, που έχουν φτάσει στα νησιά, τότε εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά το δέχομαι. Γιατί να μην μεταφερθούν αυτά τα άτομα όμως στην Υπηρετική Ελλάδα, ενώ ε, συνεχίζεται η επεξεργασία των ε, υποθέσεών τους. Γιατί να μην συμβαίνει αυτό. Για μένα, αλλά και ευρύτερα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώ, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να πούμε αν ένα άτομο έχει καταγραφεί μετά την 31η Μαρτίου στα νησιά, έχουν αποσταλεί τα δεκαλικά αποτυπώματα στην Τουρκία, μπορεί να το αυτοποιηθεί λοιπόν το άτομο. Βεβαίω για μα ε, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα θα μας διευκόλυνε ιδιαίτερος. Όμως, ε, πώ έχουν τα πράγματα σήμερα. Αυτά τα άτομα δεν μπορούν να επιστραφούν στην Τουρκία. Μετά, μπορούμε να κάνουμε διαφορετική αξιολόγηση. Να πούμε, όπω και να έχει, εμεί θα του μεταφέρουμε στην υπηρετική Ελλάδα. Και αυτό είναι μια θέση που μπορεί να υποστηρίξει κάποιο. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά αυτό υπονομεύει την κοινή δήλωση με την Τουρκία. Γιατί μετά και η Τουρκία μπορεί να πει, ή μάλλον συγγνώμη, ένα μετανάστη μπορεί να πει, ε, φτάνω στα νησιά, περνάω αρκετά γρήγορα στην ε, υπηρετική Ελλάδα και δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής μου στην Τουρκία. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ, κυρία Σετζεντίνη. Συγγνώμη που επανέρχομαι, κύριε Πρόεδρε, αλλά το θέμα δεν είναι πού φτάνει κάποιος μια συγκεκριμένη μέρα, αλλά κατά πόσο βρίσκεται ακόμα κάποιος στο νησί, αλλιώς δεν τον δέχεται πίσω η Τουρκία. Άρα η Τουρκία ε, υποδεικνύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πού να φιλοξενεί τα άτομα μέχρι να επιστραφούν. Δεν λέω ότι πρέπει να το αγνοήσουμε αυτό, δεν υπονοώ κάτι τέτοιο. Απλώς θέλω να κατανοήσω γιατί δεν τους μεταφέρουμε. Αν καταγράψουμε το γεγονός ότι φτάνουν σε ένα νησί πριν ή μετά από μια μερομηνία. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά προσθέτω ότι βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την ε, Τουρκία και συνεχίζονται αυτές οι επαφές και θέλουμε να δούμε ακριβώ αυτό. Αν θα μπορούσαμε αυτά τα άτομα να τα φέρουμε στην υπηρετική Ελλάδα και μετά να του επιστρέψουμε. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Μετά. Γιατί είναι τόσο χαμηλός ο αριθμός των ε, επανεγκαταστάσεων. Ίσως ο συνάδελφος θέλει να πει κάτι. Το μόνο σημαντικό είναι να κάνουμε διάκριση μεταξύ του κανόνα ένας προς έναν και του άλλου τμήματος του καθεστώτος επανακατάστασης. Το πρώτο τμήμα λοιπόν είναι το ένας προς έναν, που είναι ο αριθμός που αναφέρατε. Όμως είπε ο κύριος Ράιον ότι υπάρχουν και άλλες επανακαταστάσεις. Όμως να το σχολιάσω ο ίδιος. Λοιπόν, ε, εδώ συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ε, διαβίωσης ε, και φιλοξενίας ε, των μεταναστών. Εξήγησα, ελπίζω, πού είναι τα προβλήματα, η στενοπή. Δεν είναι ότι δεν έχουμε τα χρήματα, την ενέργεια, τη βούληση. Δεν έχουμε χώρο. Αν έχουμε υπερτιμήσει τον αριθμό των επανακαταστάσεων, εδώ επανερχόμαστε στον αντίκτυπο της συμφωνίας με την Τουρκία. Είχαμε τον αριθμό των 6.000 επανακαταστάσεων για την Ελλάδα. Όταν το προσδιορίσαμε αυτό, ήταν πριν από τη συμφωνία με την Τουρκία. Στη συνέχεια, έχει μειωθεί ο αριθμός των αφήξεων. Επομένως, έχει μειωθεί δραστικά και ο αριθμός ε, των επιλέξιμων σε επανεγκατάσταση. Τώρα. Εξαιρετικά σημαντικό το θέμα του συντονισμού. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Πρόκειται για κράτος μόνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την οργάνωση, όλα αυτά πρέπει να γίνονται μέσω συντονισμού. Και εμείς ελπίζουμε οι ίδιες οι αρχές, προτιμούμε μάλλον οι ίδιες οι αρχές να ε, το αναλαμβάνουν. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξουμε την Ελλάδα σε αυτό το εγχείρημα. Και η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ διαβουλεύεται και με τους εταίρους της και με, τις, ε, με το Υπουργείο Μετανάστευσης, αλλά και από πλευράς μας προσπαθούμε να στηρίξουμε κατά το δυνατόν αυτή τη διαδικασία. Με μια εύλογη κατανομή και επιμερισμό εργασιών, Υπάρχει και ειδική υπηρεσία ε, για, την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν ασχολούμαι εγώ απευθείας. Τώρα, κατά πόσο μπορούμε να δεχθούμε τη μεταφορά ανθρώπων σε ε, εργοστάσια χωρίς θέρμανση. Σαφώς και δεν είναι αυτό που θέλουμε. Τι συνέβη τις περασμένες εβδομάδες. Προσπαθήσαμε πριν από μερικούς μήνες είχαμε χιλιάδες ανθρώπους στην Ιδωμένη. Αρχικά μεταφέρθηκαν υπό πολλές επικρίσεις σε άλλους χώρους, αποθήκες κτλ. Τώρα όπου μπορούμε βελτιώνουμε τις συνθήκες σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπου δεν είναι αυτό δυνατόν, τους μεταφέρουμε αλλού. Αυτή είναι η δικασία που ακολουθείτε. Και από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, έχουμε ακόμα περίπου 700 ανθρώπους, τουλάχιστον χθες έτσι ήταν. που καταβάλλονται προσπάθειες να μεταφερθούν σε καλύτερους χώρους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πιέσεις προς το ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθελψης, το οποίο ισχύει. Και η Γενική Διεύθυνση Home έχει παράσχει ε, κατεπίγουσα βοήθεια προς ε, ε, το σύστημα υγείας. Αν τα κρατημέλη κάνουν αρκετά για την μετεγκατάσταση. Δεν θέλω και πάλι, φοβάμαι να χρησιμοποιήσω διπλωματικούς όρους, γιατί με κατακρίνατε πριν αλλά κάνουν περισσότερα από ό,τι έκαναν πριν, όπως είπε και ο κύριος Ράιαν. Τώρα έχουμε τους τελευταίους μήνες περίπου χίλιες ε, μετακαταστάσεις το μήνα. Βεβαίως και θέλουμε να αυξηθεί αυτός ο αριθμός στους 2.000 και τα 3.000 τον Απρίλιο. Το έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι αυτό εντάσσεται και στο κοινό σχέδιο δράση που έχει υιοθετηθεί και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υποθέτω λοιπόν ότι και τα κράτη-μέλη θα καταβάλουν προσπάθειες ε, για την ολοποίησή του. Αν αυτό τώρα συνδέεται με την... Αν μάλλον η διαδικασία ε, αποδοχής ε, παρεμποδίζει άλλες ε, συνθήκες για την οικογενειακή επανένωση. Στην πράξη αυτό βλέπουμε. Ότι δηλαδή δεν παρεμποδίζει η διαδικασία επανένωση ή ε, την ε, εξέταση τη αίτηση. Δεν γνωρίζω τι ισχύει με τις ε, συμφωνίες με τη Λιβύη, αν πρέπει να το πράξουμε ή όχι, δεν θα σχολιάσω. Οι μετανάστες βρίσκουν νέες οδούς προς την Ευρώπη, αναμφίβολα, έχουν φαντασία οι άνθρωποι. αλλά τουλάχιστον ως προς την ε, Ανατολική Μεσογειακή Οδό, προς την Ελλάδα, ε, βλέπουμε πολύ λίγες ενδείξεις για συνέχιση αυτής της ε, ροής. Είδαμε ότι από τις 900.000 έχουμε πέσει. Στην κεντρική Μεσόγειο έχει αυξηθεί κατά 26.000. Αλλά έτσι κι αλλιώς μιλάμε για διαφορετικές ομάδες μεταναστών. Σταματώ εδώ έχουν τρένα οι βουλευτές μου να πάρουν ε, και αεροπλάνα και τέτοια. Βέβαια καλά κάνατε και είπατε για κάποιες λεπτομέρειες. Εσείς τώρα. Εγώ νομίζω ότι ο συνάδελφός μου κάλυψε τις περισσότερες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Δεν νομίζω να μείνουν πολλές. Μία ερώτηση ήταν γιατί θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον στόχο της επίτευξης των μετεγκαταστάσεων στους αριθμούς του Σεπτεμβρίου 2015. Ερώτηση κυρίας Πόστ και του κύριου Λέναρς. Μήπως υπερεκτιμήσαμε τον αριθμό των ε, προσώπων που είναι δυνατόν να μετεγκατασταθούν. Νομίζω το σωστό είναι να πει κανείς ότι τον Σεπτέμβριο 2015 το Συμβούλιο ανέλαβε μια δέσμευση με τα βλέμματα στραμμένα προς τα μπρος για τους αριθμούς των προσώπων που είναι δυνατόν να μετεγκατασταθούν. Μαθηματικά ε, εάν δεν γεμίσετε πλήρω το μπουκάλι δεν μπορείτε, το ε, ποτήρι δεν μπορείτε και να το πιείτε το περιεχόμενο. Αυτό εξηγεί και για ποιο λόγο η Κομισιόν κάπως ε, μετρίασε ή μάλλον ε, μετέτρεψε τους στόχους. Προσαρμόζουμε τους στόχους δηλαδή τώρα σε ό,τι αφορά τον αριθμό ατόμων που θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να μετρικασταθούν όσο οι εισρωές, οι τρέχουσες εισρωές παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Νομίζουμε ότι αυτό ε, είναι λογικό. Κάποιες ερωτήσεις τέθηκαν επίσης πάλι νομίζω την κυρία Πόστ και τον κύριο με, το, με την έννοια πως συμφιλιώνουμε τις προφανώς ο πρόεδρος διακόπτη. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε κάποια παρανόηση υπήρξε. Ο πρόεδρος διευκρινίζει την παρανόηση. Πώς συμφιλιώνουμε λοιπόν το γεγονός ότι προφανώς έχουμε ελληματικές εγκαταστάσεις υποδοχής ο τρόπος με τον οποίο συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να ξαναρχίσουν οι μεταφορές Δουβλίνου. Εξειδικεύει στο κείμενο της Επιτροπή ότι οι εξασφαλίσεις αυτές, οι διασφαλίσεις αν θέλετε, πρέπει να αναφέρονται και στα καταλήματα τα οποία θα υποδεχτούν τα πρόσωπα αυτά. Η Ελλάδα δηλαδή θα πρέπει να δώσει μια εγγύηση ότι το πρόσωπο που θα μεταφερθεί θα έχει μια θέση σε μια κατάλληλη δομή υποδοχής η οποία θα ανταποκρίνεται σε κάποιες προδιαγραφές. Κάτι το οποίο φαίνεται να είναι αντιφατικό, ίσως στην ουσία να μην είναι. Αλλά να είναι υλοποιήσιμο και μάλιστα με τρόπο σύμμορφο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μία ερώτηση γενικού χαρακτήρα που θέσατε και την οποία πίντησε ο Μάρτιν εν μέρη γιατί δηλαδή οι αριθμοί των επανεγκαταστάσεων είναι τόσο χαμηλή γενικά Το ερώτημα αυτό τίθεται μέσα σε διαφορετικά πλαίσια, σε πολλά και διαφορετικά πλαίσια δηλαδή. Είναι δύσκολο να απαντηθεί, είναι περίπλοκο να απαντηθεί, αλλά προσπαθώντας να απλοποιήσω μια πρώτη απάντηση, Ίσως η καλύτερη απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι να πει κανείς ότι οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκαν λιγότερο γενναιόδορες σε ό,τι αφορά την ε, χορήγηση θέσεων επανεκατάστασης από άλλα μέρη του βιομηχανοποιημένου κόσμου. Λόγω του γεγονότος απλώς ότι οι αιτήσει ασύλου προέρχονται από αφήξεις στην βάση βέβαια της γεωγραφικής θέσης Τη Ευρώπη, Αν τα συγκρίνετε για παράδειγμα με τι Ηνωμένε Πολιτείε ή με την Αυστραλία που έχουν την πολυτέλεια των εισαγωγικών να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρούν τις υποχρώσεις τους απέναντι σε πρόσφυγες. Και πιο πολλοί από τους πρόσφυγες έρχονται μετά από, ή μέσα στα πλαίσια επανεγκαταστάσεων. Νομίζω ότι καλύπτω λίγο πολύ όλες τις ερωτήσεις που μου θέσατε ή μας θέσατε και που δεν είχαν ήδη απαντηθεί από τον φίλο Βερβέη. Α, εσείς είχατε. Ναι, ρώτησα για τα λεφτά, λέει η κυρία Λάμπερτ. Αν δηλαδή είστε ήσυχο ότι όντως γνωρίζετε πού πάνε τα χρήματα. Ναι, πράγματι. Οφείλω να πω σχετικά με το ερώτημά σας ότι δεν έχω την αναγκαία τεχνογνωσία και background για να σας απαντήσω πλήρως την ερώτηση σας. Προτιμώ να μην σας απαντήσω λοιπόν. μπορώ να φέρω τη γραμματεία σας σε επαφή με τις οικονομικές μας υπηρεσίες, εκτός αν ο κύριος Βερβέη δεν είμαι βέβαια εγώ αυτός που εγκρίνει τις δαπάνες, λέει ο κύριος Βερβέη, αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει ένας αριθμός διασφαλίσεων το ΕΚΟ έχει και ένα μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται και έχει εφαρμοστεί και αλλού που περνά μέσα από έμπιστους εταίρους η ροή του χρήματος που οφείλουν να συμμορφώνονται σε ορισμένα πρότυπα λογιστικά και άλλα. Ο ΕΚΟ λοιπόν ακολουθεί την οδό αυτών των διασφαλίσεων και η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών, home δηλαδή, έχει τα σχετικά πρότυπα. Δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο σε αυτά, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαφώς όπως κάθε ευρωπαϊκή δαπάνη ε, πρέπει να υπάρχει πλήρης λογοδοσία απόδοση λογαριασμών αν θέλετε αλλά νομίζω ότι είναι κάπως πρόημο να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση τώρα Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε επικαλύψεις δαπανών. Αλλά έχετε δίκιο που τονίζετε το σημαντικό αυτό παράγοντα. Όπως είπα, ίσως δεν είμαι απόλυτα αρμόδιος να σας απαντήσω. Μπορεί το οικονομικό μας τμήμα να σας δώσει μια απάντηση όταν θα έχει προχωρήσει προσπάθειας προσπάθεια. Ένα πρόσθετο θέμα, κύριε Ράιαν, να απαντήσω σε μια ερώτηση που έθεσε ο κύριος Λέναρτς σχετικά με το ότι θα πρέπει να επιτρέπονται οι μεταφορές του Δουβλίνου μόνο υπέρ των χωρών μελών εκείνων που ταυτόχρονα προσφέρουν και θέσεις για επανεγκατάσταση. Πράγματι, ε, είναι μια ελκυστική ιδέα, αντιλαμβάνομαι ποια μπορεί να είναι η ελκυστικότητα που ασκεί, αλλά η απάντηση που θα μας δώσει, μας δώσει η Επιτροπή είναι ότι οι νομικές υποχρώσεις δεν είναι, ε, πώς να πω, διαπραγματευτές. Δεν είναι διαπραγματεύσιμες, ε, ζητή συγγνώμη για ε, δεν είναι διαπραγματεύσιμες, είναι νομικές υποχρώσεις σε ό,τι αφορά την επανεγκατάσταση. Και βεβαίω υπάρχει και υποχρέωση για την Ελλάδα να σέβεται την ισχύ του δικαίου. Και όλα αυτά πρέπει να κινηθεί μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Πριν να βιαστείτε, να σηκωθείτε και όλοι θέλετε να προλάβετε τα διάφορα μέσα μεταφοράς. Κανείς από τους αρμόδιους ηγητές δεν ήταν παρόν λόγω του χρονοδιαγράμματος της ε, σχετικής συζήτησης. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήσασταν παρούσες εδώ και θέσατε τα ε, θέματα αυτά και μάλιστα με αρκετή έμφαση και με κάποια ε, πώς να πω, ε, συναισθηματική φόρτιση που είναι απόλυτα κατανοητή, γιατί μιλούμε για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων εδώ. Και είναι αυτονόητο. Ευχαριστώ λοιπόν τα μέλη που έθεσαν τα θέματα. Ευχαριστώ και τους δυο σας, εσάς αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι χρειαζόμαστε ε, διαρκή αναφορά εκ μέρους σας Βεβαίως υπάρχουν σαφείς αποκλήσεις αποφάσεων και μεταξύ σας και μεταξύ των μελών μας. Η δική μου προτεραιότητα πάντως είναι, είναι να διατηρήσουμε ε, τον, ε, τον διάλογο αυτό και να συνεχίσουμε να συζητούμε τα βασικά από αυτά τα πρακτικά θέματα να διατηρηθεί η συζήτηση αυτή γιατί στρέφεται γύρω από πολύ σημαντικά θέματα ανθρωπιστικά θέματα. Ευχαριστώ λοιπόν που παραμείνατε εδώ. Σας ευχαριστώ και πάλι και τους δυο σας. Η επόμενη συνάντησή μας την 31η Πρώτου θα είναι καταστατική. Δηλαδή θα συγκροτήσουμε εκ νέου την ε, Επιτροπή μας. Άρα να είστε εδώ. Δεν μπορείτε να λείψετε. 31 πρώτου. Ευχαριστώ όλους και όλους που μείνατε μέχρι του τέλους. Για τα διάφορα τίποτε. Λίγη συνεδρίαση.